I hope that everybody had a nice Ελπίζω να ξεκουραστήκατε όλοι κατά τη μεσημεριανή διακοπή, έτσι ε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω σε εσά για την ετήσια έκθεση όσον αφορά τι δραστηριότητε του διαμεσολαβητή για τη χρονιά που μα πέρασε. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία που είχαμε για αυτή την έκθεση. Και κατάφερα να δεχτώ τις περισσότερες ε, τροπολογίες που κατέθεσαν οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, μπορείτε αυτό να το δείτε στο σχέδιο της έκθεσης που σας ε, κατατέθηκε. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω το εξής γεγονός, ότι η έκθεση της κυρίας Ρέγη της Ευρωπαίας Διαμεσολαβητού ήταν ιδιαίτερα προσιτή και φιλική και θα ήθελα να φέρω δύο θέματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα. Προτείνω λοιπόν ότι αντί να αναφέρονται οι χαρακτηριστικές 100 αναφορές, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία στις ετήσιες εκθέσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και μία σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα έτη και με ευκολία μάλιστα. Και αυτό θα διευκολύνει να διαπιστώσουμε τάσεις που επικρατούν στο επιτρεπτό των αναφορών ή όχι. Και με βάση τις πληροφορίες που έλαβα, αυτό ελήφθη υπόψη στις ε, εργασίες και στην έκθεση του 2014. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Διαμεσολαβητή για το ότι έλαβε υπόψη σε αυτή την παρατήρησή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένας πολύ χρήσιμος οδηγός στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Χρηστή διαχείριση και πρακτική, οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013. Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε αποκλειστικά και μόνο στα αγγλικά. Εξ όσων γνωρίζω υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι οικονομικοί περιορισμοί για τη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες, όμως εδώ πρόκειται για μια ε, επίσημη έκθεση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο, άρα θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το τι έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και έχει κοστίσει 5.000 ευρώ. Άρα δηλαδή το ποσό είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η έκθεση να μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες. Επίσης, ορισμένοι σκιώδεις συζητητές ανέφεραν ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι ειδικέ εκθέσεις, κυρίως αυτή που αφορά τη Frontex. Και όσον αφορά την πρόταση για την, ε, ε, για την έκθεση αυτή που υποβάλλεται στην Επιτροπή Αναφορών, εξακολουθούμε να περιμένουμε την, Επιτροπή, την διάσκεψη των Προέδρων γιατί έτσι και αλλιώς θα μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Ας μην μιλήσουμε λοιπόν δυο φορές για το ίδιο πράγμα και μια άλλη τεχνική παρατήρηση που αφορά τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Είχα προβλέψει μια τέτοια συνάντηση καταρχήν για την επόμενη εβδομάδα. Όμως γνωρίζω ότι οι πράσινοι και η Ηνωμένοι Αριστερά θα έχουν πρόβλημα με συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν οι συνάδελφοί μας να ενημερώσουν τη γραμματεία για το πότε είναι διαθέσιμη εμείς προτείνουμε την Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 10 ή από τις 10 μέχρι τις 11. Θα ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε την έκθεση αυτή να την παρουσιάσουμε μετά από ε, διαβουλεύσεις με όλους. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, το λόγο έχουν οι συνάδελφοι Γιούλια Ρέντα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική συνεργασία, ε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το ότι υπήρχε πίεση χρόνου και θα έχουμε περιορισμένο χρόνο κατά τις επόμενες εβδομάδες. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, αρκετά ικανοποιημένοι με την έκθεση και επίσης ε, εκτιμούμε το γεγονός ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι αριθμοί στην έκθεση. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελα να συμπεριλαμβάνεται και αυτό, πέρα από αυτά που ήδη συζητήσαμε, και αυτό το θέμα είναι η φύση της ειδική ε, έκθεσης. Δηλαδή η διαμεσολαβητής έχει εδώ ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ένα του και στην ειδική έκθεση αναφέρεται ότι η διαμεσολαβητής ε, θέλει την κοινοβουλευτική υποστήριξη για να ε, συνεχίσει αυτήν την έκθεση για τη Frontex. Θεωρώ λοιπόν ότι παρότι η έκθεση είναι ιδιαίτερα θετική όσον αφορά τη δουλειά της και επίσης ε, εκτιμούμε το γεγονός ότι προσπάθησε να ε, εξετάσει λίγο τις περιπτώσεις της κακοδιαχείρισης. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να μην αναφέρονται μόνο αυτά τα γενικά λόγια, αλλά να αποδοθεί και ιδιαίτερη σημασία στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Εκ μέρου λοιπόν των Πρασίνων θα ήθελα να πω ότι επιθυμούμε να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση του Κοινοβουλίου στην έκθεση αυτή, δηλαδή ότι θα συντάξουμε μια δική μας έκθεση πρωτοβουλίας για την ειδική έκθεση, ακόμα και αν κάποιες ομάδες διαφωνούν με τα συμπεράσματα αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης. Όμως, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, έτσι ώστε η ειδική έκθεση να καταστεί πράγματι ένα ατού στα χέρια της διαμεσολαβητού και με την έννοια ότι θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι αυτή είναι ε, μια δυνατότητα έσχατης καταφυγής, ένα ατού όπως είπαμε που έχει στα χέρια της. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να υπάρχει έτσι μια τέτοια ηχηρή αναφορά στην έκθεση. Και είπατε βέβαια και εσείς ότι το κόστος της ε, μετάφρασης σε όλες τις γλώσσες ε, είναι υψηλό. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει τα έγγραφα ε, που απευθύνονται στην κοινή γνώμη, αυτά θα πρέπει να μεταφράζονται. Έτσι ώστε να μπορούν όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες να έρχονται σε επαφή με τη δουλειά της ε, διαμεσολαβητού. Και βεβαίως και θα πρέπει να δούμε και τα κονδύλια που διατίθενται στη διαμεσολαβητή για να μπορεί και εκείνη να εκτελεί τα καθήκοντά της με το σωστό τρόπο, που είναι πάρα πολλά και εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να ανακεφαλαίωσω λιγάκι τι συζητήσαμε σήμερα το πρωί στις συνεδρίες των συντονιστών. Αποφασίσαμε ήδη ότι αυτό το θέμα θα έχει πρώτη προτεραιότητα η Επιτροπή Αναφορών σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθερίων που είναι η νομοθετική επιτροπή είναι αυτή που θα κάνει τη δουλειά ε, σε σχέση με την έκθεση Frontex ε, βάσει του άρθρου 55. Δεν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτή την έκθεση. Η Μπέα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα για την ταχύτητα και τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο εκπώνησε αυτή την έκθεση και θέλω να χαιρετήσω και την ε, καλή του διάθεση. Δέχτηκε να συμπεριλάβει τροπολογίες του Άλντε και σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφος των Πρασίνων πρέπει και εγώ να τονίσω ότι η έκθεση αυτή είναι σημαντικό εργαλείο για να καταστήσουμε σαφές ότι όπως ε, θα μπορούσε να πούν και όσοι να μπορούσε να πει και κάποιος ε, που του ε, αρέσει η μυθολογία η αντιμετώπιση μας είναι διπρόσωπη σαν τον Ιαννό της μυθολογίας από τη μία πρέπει να στηρίξουμε τη δραστηριότητα της διαμεσολαβήτριας γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά τα λόγια και γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω όταν καταλήξουμε στην τελική εκδοχή πέρα από τη χρήση εκφράσεων όπως ε, χαιρετίζω, σημειώνω και τέτοια να πούμε ότι στηρίζουμε, ενισχύουμε, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες, δράσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην έκθεση για τις επιπτώσεις, ε, τη σχετικότητα και την ορατότητα της δραστηριότητας. Επίσης έχουμε και τις ε, διαβουλεύσεις που έχουν γίνει για τη διαφάνεια, η οποία μόλις έκλεισε και περιμένουμε τις, ε, τα απορίσματα για τη Συμφωνία Εμπορίου με τις Ηνωμένε Πολιτείες και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις περιστρεφόμενες πόρτες. Δηλαδή με το πώς κάποιοι που συνταξιοδοτούνται παίρνουν μετά καλές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών που είναι όργανα κλειδιά να αποδείξουμε ότι δεσμευόμεθα και οι δύο για να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Σμίτση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γουαλένσα, που εξεπώνησε μια πολύ καλή έκθεση και με χαρά διαπιστώνω ότι πολλές από τις τροπολογίες ε, που είχαν προτείνει οι σοσιαλιστές και ο Σκιώδης, ο δικός μας, συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Είναι σημαντικό για μας να συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά, όπως ακριβώς και πρόκειται να γίνει, για να συμπεριληφθούν και άλλες τροπολογίες που επίσης είναι σημαντικές ε, στο τελικό κείμενο πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει αναγκαία σημασία στους πολίτες μας, να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, να ξέρουν τι κάνει ο διαμεσολαβητής, τι δραστηριότητες ε, ε, εκτελεί ο διαμεσολαβητής. Πολλοί δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τι κάνει ο διαμεσολαβητής. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δοθεί αυτή η πληροφόρηση, γιατί αλλιώ ε, στην ουσία είναι διάκριση για του πολίτε αυτού που δεν έχουν ε, καμία ενημέρωση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το παραδεκτό και το απαράδεκτο. Γιατί υπάρχουν τόσες ε, διαμαρτυρίες για κάποια θέματα που δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Η μέση διάρκεια εξέταση είναι 18 λεπτά. Είναι πολύ 18 λεπτά να περιμένει κανείς μέχρι να καταλάβουν οι πολίτες ότι επιτέλους έχει αντιμετωπιστεί το θέμα τους. Αυτό συνδέεται βεβαίως και με έλλειψη προσωπικού ενδεχομένως, αλλά και με έλλειψη επαρκούς διάθεσης να ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι τη σημασία αυτής της πλευράς του θέματος. Και συμφωνώ με τον κύριο Γουαλένσα ότι δεν πρέπει εδώ να συζητήσουμε το θέμα Frontex. Υπάρχουν άλλα πλαίσια που μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και πρέπει περαιτέρω να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την εργασία τη διαμεσολαβήτρια. Είναι πολύ σημαντικό, παραλαμβάνω, για του πολίτε και τονίζω επίση ότι θα θέλαμε να έχουμε μετάφραση αυτή τη έκθεση. Βεβαίω, κοστίζει η μετάφραση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση και τι υπηρεσίε που παρέχουμε στου πολίτε, που πρέπει να μπορούν ακριβώ να έχουν την ενημέρωση αυτή στη γλώσσα του. Και τέλο, να ευχαριστήσω την ε, Emily Riley την ε, διαμεσολαβήτρια που έδειξε πολύ θετική διάθεση και κατάφερε να υπάρχει σωστή σύνδεση μεταξύ ημών και αυτής. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα η Ελεονόρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τα θετικά σχόλια των συναδέλφων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που μας παρουσίασε. Εμείς ως ομάδα ε, θέλουμε απλώς ε, να προσθέσουμε μερικά στοιχεία στη δουλειά που έχει γίνει ήδη γίνει, να προσθέσουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις, παραδείγματος χάρη τη δυνατότητα να υπάρξει βελτίωση στην επικοινωνία μας με τους πολίτες, να προβάλλεται περισσότερο ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και αυτό μπορεί να γίνει και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς αυτό μπορεί να γίνει για να ενθαρρύνουμε περισσότερο τους ε, πολίτες να καταφεύγουν στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Κατά τα άλλα υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο του διαμεσολαβητή, πως ε, ο ρόλος αυτός ε, μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη από πλευράς πολιτών, κάτι το οποίο δυστυχώς σήμερα φθήνει όσον αφορά τις ε, τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί αυτό είναι συνέπεια της πολιτικής λιτότητας η οποία πλήττει κυρίως τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Εμείς λοιπόν προτείναμε να υπάρξει ένα σχόλιο προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης θέλω να προσθέσω ότι θα επιθυμούσαμε στην παράγραφο υπαριθμών 10 να προτείνουμε το εξής, να υπάρξει αναδιατύπωση του κειμένου δηλαδή με την εξής έννοια να επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για το ότι υπάρχουν, διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των αναφορών οι οποίες υποβάλλονται και αφορούν τις, τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της τάσης για να υπάρξει βελτίωση. Και κατά τα άλλα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τη δουλειά που μας παρουσίασε ο συγητής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Now, Mr. Marias, please. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή τον κύριο Βαλέσα διότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην έκθεσή του αυτό νομίζω το ομολογούν όλοι οι συνάδελφοι και πράγματι η έκθεση έχει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι άρτια θα έλεγα από τεχνικής απόψεως και νομίζω ότι έχει θίξει τα κυριότερα ζητήματα. Οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις των άλλων εισηγητών είναι σημαντικές και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε ένα ζήτημα σημαντικό το οποίο επηρεάζει ε, και τη λειτουργία ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ε, και βεβαίως στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτό έχει σχέση με τα αποκαλούμενα μνημόνια, δηλαδή αυτά τα θεσμικά υβρίδια μέσα από τα οποία υπήρξε μια συνεχής παρέμβαση της Τρόικας στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κρατών μελών και επηρέασε την καθημερινή ζωή, το επίπεδο το βιωτικό των λαών της Ευρώπης και κυρίως βεβαίως όσων χωρών μπήκαν σε μνημόνια, τους οποίους φτωχοποίησε και έτσι παραβιάστηκαν και τα δικαιώματά τους. Εδώ λοιπόν έχουμε τέσσερα σημεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, ότι η ίδια η λιτότητα οδηγεί σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει διαπιστώσει ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο κύριος Μούζνιετς του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάπως αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μέσα στην έκθεση. Θα υποβάλουμε συγκεκριμένες τροπολογίες προς τον συνάδελφο τον κύριο Βαλέσα για να διευκολύνουμε τις ε, παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε ούτως ώστε να συμπεριληφθούν. Το δεύτερο έχει σχέση με το παραδεκτό. Διότι το παραδεκτό μιας αναφοράς επίσης εξαρτάται υποτίθεται από το αν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμω, μέσω της Τρόικας αυτό που έγινε είναι να παρεμβαίνει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα τα οποία παλαιότερα ήταν εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά στην πράξη η παρέμβαση αυτή επηρεάζει τα δικαιώματα των πολιτών. Άρα το θέμα του παραδεκτού τροποποιείται πιστεύω σε μεγάλο βαθμό λόγω των μνημονίων τα οποία λειτουργήσαν επί αρκετά χρόνια σε χώρες που βρέθηκαν σε μνημόνιο. Το τρίτο θέμα και πιο σημαντικό είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Και εδώ έρχεται να παίξει ρόλο ο διαμεσολαβητής. Θα θυμόσαστε είχα θέσει αυτό το ζήτημα στην ε, διαμεσολαβήτρια η οποία ήταν παρούσα και της είχα πει ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της, εντός της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μια πλευρά υποτίθεται ότι είναι ο θεσμός που προστατεύει το ευρωπαϊκό συμφέρον, το κοινό συμφέρον. Και από την άλλη είναι ο εκπρόσωπος των δανειστών στις χώρες που βρίσκονται σε μνημόνια. Αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων. Δεν το λέω εγώ. Υπάρχει ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ψηφιστεί φέτος τον Μάρτιο και τα λέει. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του διαμεσολαβητή στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να αναζητηθεί και άρα θα πρέξει, πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Και θυμάμαι την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια που είπε ότι αυτό το θεωρεί σημαντικό και θα το εξετάσει. Και από εκεί και πέρα μπαίνει το ζήτημα πώς θα εκδηλωθεί αυτή η παρέμβασή της, δηλαδή θα εξετάσει και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι είναι. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Τρόικας και ταυτόχρονα ο θεσμός που προστατεύει την νομισματική πολιτική και ταυτόχρονα ο δανειστής συγκεκριμένων κρατών μια και έχει αγοράσει ομόλογα της Ελλάδας της Ιταλίας, της Ισπανίας κλπ. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και θα καταθέσουμε κύριε Βαλέσα ε, δύο τροπολογίες στο ζήτημα αυτό. Θα μιλήσουμε μαζί σας, ούτω ώστε να μπορέσουμε να θίξουμε αυτά τα ζητήματα μέσα στην έκθεση. Γιατί αυτά τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Κατά τα υπόλοιπα, η συμφωνία μας υπάρχει στα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Now I'll give the floor to, to Mrs. Auken, please. Η κυρία Auken τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω την παράδοσή μου και θα μιλήσω και πάλι δανέζικα όπως κάνω συνήθως. Μία ερώτηση έχω που έχει να κάνει με το διαμεσολαβητή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βαλένσα για το εξαίρετο έργο του. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Όμως μια πληροφορία ότι θα κλείσει η υπόθεση αυτή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το ETIP. Ήδη το ακούσαμε, αλλά σήμερα μια εφημερίδα στη Δανία έχει ένα μεγάλο άρθρο για το κόστος της συμφωνίας αυτής που έρχεται σε αντίφαση με αυτά που μας έχει πει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική πτυχή της συμφωνίας αυτής, την απασχόληση κλπ. Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα για πιο συγκεκριμένα τι υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Και γι' αυτό πολύ χαρικά όταν η ίδια Μεσολαβητή ζήτησε μεγαλύτερο άνοιγμα όσον αφορά την εντολή πιστεύω και εγώ ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη εντολή για το τι βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Συζητάμε για το SDN, αυτό το ειδικό δικαστήριο διατησίας ουσιαστικά που λέμε ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά εμπόδια το SDS. αν τελικά πραγματοποιηθεί έτσι όπως προβλέπετε. Πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες μας και χρειαζόμαστε ανοιχτό πνεύμα για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος, ε, κύριε Χάσικαμπ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ρόλος του Ευρωπαίου Μεσολαβητή. Η αλήθεια είναι ότι γεννήσαμε πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και είναι καλό που βλέπουμε ότι ακούγονται οι πολίτες πια. Έχω βέβαια κάποια, κάποιους δισταγμούς όσον αφορά το τι γίνεται με τις συστάσεις. 80% ακούσαμε ότι είναι οι αποφάσεις ποιες από αυτές τις συστάσεις τελικά όντως ε, ακολουθούνται και δυστυχώς το ποσοστό δεν είναι μεγάλο. 80% των συστάσεων δεν ακολουθούνται τελικά από τα όργανα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να βαρύνουν περισσότερο οι συστάσεις του διαμεσολαβητή. Γι' αυτό και θα υποβάλω σχετική τροπολογία. Ωραία, εδώ ολοκληρώνεται το κατάλογο ομιλητών που είχα, λέει η Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ, αλλά δεν επιθυμεί να πάρει το λόγο σε αυτό το στάδιο. Οπότε θα σας δώσω το λόγο σε εσά πάλι κύριε Βαλέσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή, ποιος είναι ο ρόλος του και τα καθήκοντά του και να μην το ξεχνάμε αυτό. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο το μεσημέρι στις 12. Συνεπώς, περιμένω ότι άλλες τροπολογίες έχετε να μου τις στείλετε έγκαιρα και μετά θα καθίσουμε κάτω με τους σκιώδες εισηγητές να τις συζητήσουμε και σίγουρα θα καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε και μόλι ο εισηγητής, ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο 12 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Η ακρόαση με τη διαμεσολαβητή θα λάβει χώρα επίση στι 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Σας ενημερώνω επίσης και το εξής. Θα θυμόσαστε ότι στείλαμε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που του ζητούσαμε να δημοσιοποιήσει με πλήρη διαφάνεια όλες τις υπογραφές των Ευρωβουλευτών. Πήγε προς την κατεύθυνση που του ζητάμε, αλλά όχι πλήρως. Τι έκανε. Έδωσε τις οι υπογραφές, αλλά σε μια συγκεκριμένη αίθουσα πάνω. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και μου έφτασε ένα σχόλιο που λέει, ε, ας πούμε τότε στον πρόεδρο να πάει να τις φωτογραφίσει και να τις ε, φορτώσουμε, να τις έχουμε όλοι. Πράγματι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να δώσουμε συνέχεια. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε στην αίθουσα αυτή, να διαβάσετε τις υπογραφές και να ενημερωθείτε με τη μέθοδο αυτή. Δεν είναι βέβαια αυτό που είχαμε εμείς υπόψη μας όταν στείλαμε την επιστολή, με την οποία ζητούσαμε πλήρη διαφάνεια, αλλά είναι αν μη τι άλλο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία, ολοκληρώσαμε έτσι το σημείο 11 και περνάμε στις αναφορές μας και πάλι. Σημείο 12. Αναφορά 0873 του 2013 του Κλοντ cost. Είναι εδώ για τα θέματα πλημμυρών στη Γαλλία. Είναι εδώ ο κύριος Κώστα. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Λίγα λεπτά χρειάζομαι μόνο. Κυρία Πρόεδρε, Τέσσερι νεκροί μετά από τις καταρακτώδεις βροχέ τη ΕΒΕΝ το Σεπτέμβριο του 2014 στο Λακεντόκ Ρουσιών. Με βροχέ μέχρι 400 mm. Έρευνα, υποτροπή, ανάλυση αιτιών είναι πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στην οδηγία που έχει να κάνει με τη διαχείριση των κινδύνων για πλημμύρες. Μπορούμε να φανταστούμε μια πυρηνική καταστροφή χωρίς να υπάρξει έρευνα, χωρίς να γίνει μελέτη των αιτιών για να αποφύγουμε την επανάληψη. Ε, εδώ με τις πλημμύρες αυτό ακριβώς έγινε. Υπάρχει η οδηγία 2007-60 που λέει ότι οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να αποφευχθούν αλλά αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνουμε αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις ε, πλημμύρες επειδή ακριβώς δεν κάνουν τίποτα για να τις αποφύγουν. Όλα αυτά όμως θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί ή τουλάχιστον να μειωθούν οι επιπτώσεις με την οδηγία που έχει να κάνει με τις πλημμύρες ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία του πληθυσμού στην Ευρώπη γνωρίζοντας τους κινδύνους και την τήρηση των νόμων και των κανόνων που ισχύουν. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αυτό. Εγώ είχα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την, ε, ε, την αφορά 340 ε, πήγα στην Επιτροπή και με άκουσε και ο κύριος Βαρόσο. Υπάρχει λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο. Η ευθύνη της προκαταρτικής έρευνας είναι των γαλλικών αρχών στα πλαίσια της νέας οδηγίας. Είναι μια έρευνα η οποία πρέπει να καλύψει ανάλυση κινδύνων και αιτιών που προκαλούν πλημμύρες και να συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση συμμετοχής του κοινού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να την κάνει την έρευνα. Λοιπόν, από το 2007 αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε, είμαστε 2014, σε 10 χρόνια εγώ δεν θα είμαι σε θέση να ξανάρθω και να τα ξαναπώ και όλα αυτά τα εκατομμύρια των ε, Γάλλων πολιτών που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες, οι Ευρωπαίοι κτλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους βράφει στα παλιά της τα παπούτσια. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν οι πλημμύρες, ε, το νερό, η λάσπη, που αποδείχτηκαν οι κίνδυνοι μάλιστα της ρήπανσης από τη λάσπη αυτή από το σκάφος του Μέντε που τα ήλεξε όλα αυτά. Οι ακτές κινδυνεύουν, όπως έγινε στο Μπεζιέ Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν αφορούν μία χώρα, αλλά ένα σύνολο χωρών που θα υποστούν τι συνέπειες. Η Γαλλία ή κάποια άλλη χώρα δεν έχει το δικαίωμα να πει κάνω ό,τι θέλω γιατί είναι η χώρα μου και αδιαφορώ για τις συνέπειες για το περιβάλλον, γιατί 90% των πλημμυρών προκαλούνται τεχνητά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αλλού ε, γη η οποία δεν έχει αξία να γίνει γη με αξία γιατί μπορεί να χτιστεί. Είναι δράματα λοιπόν από καταστροφές που λέμε ότι είναι φυσικές, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ζητάω λοιπόν για τους Ευρωπαίους να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ασφάλεια, να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης για να αποφύγουμε τις κλιματικές καταστροφές και απαιτώ έρευνα μετά από κάθε καταστροφή με υποχρέωση να συμμετέχουν και όσοι είναι θύματα τέτοιων καταστροφών. Αυτό έχω πει και στον κύριο Παρόσο. Ζητάω επίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει τα χρήματα, τα οποία τα κονδύλια δηλαδή που πηγαίνουν στι χώρε για να γίνουν διάφορε διευθετήσει, να μην χρησιμοποιούνται για να επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά τι πλημμύρε ή για να κλείνουν οι γέφυρε από κάτω, όπω έχει συμβεί με τα έξι τόξα τη παλιά γέφυρα του Μπεζιέ. Επειδή τάχα μου γίνονται έργα για τουριστικού σκοπούς. Και αντίθετα με αυτά που λένε οι γαλλικές αρχές για τις συνέπειες της άρνησης να αφήσουμε τα νερά της βροχής να φεύγουν ελεύθερα για δεκάδες χιλιόμετρα, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ανάγκη για τον κόλπο της Γασκόνης και η προστασία των ακτών. Έχουμε καταθέσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία με την αναφορά μας αυτή. Από το 1995 λοιπόν είχαμε τους πρώτους νεκρούς από τις πλημμύρες στο Πεζιέ και από τότε προσπαθώ να διορθώσω την κατάσταση. Έχω συναντηθεί με διάφορους συνομιλητές αυτούς οι οποίοι υφίστανται τα αποτελέσματα των ε, πλημμυρών, αυτούς που κερδίζουν από χάρη, χάρη στις πλημμύρες αυτές και εκείνοι οι οποίοι με ελάχιστες εξαιρέσεις κορυδεύουν την όλη Ευχαριστώ τώρα είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάβελ Μίσιγκα, ε, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θα παρουσιάσω την άποψη της Επιτροπής για τις δύο αναφορές 873 και 943. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τον αναφέροντα για το θέμα της διαχείρισης των κινδύνων ε, πλημμύρας. Είναι πολύ σημαντική κίνδυνη, πρέπει να υπάρχει διαχείρισή των. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη χρηστή διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες με την οδηγία 60 κάθετος 2007 ε, η οποία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να δεξαγάγουν προπαρασκευαστική αποτίμηση των κινδύνων πλημμύρας και να αναπτύξουν χάρτες ε, για τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες μέχρι το τέλος, το τέλος του 2013 και μετά με βάση την χωρική κατανομή αυτών των κινδύνων και την ε, αναμενόμενη διάσταση αυτών των πλημμυρών είναι αναγκαίο οι χώρες μέλη, τα κράτη-μέλη, μέχρι τέλους του 2015 να εκπονήσουν προγράμματα αντιμετώπισης. Αυτά τα διαχειριστικά προγράμματα πρέπει να καθορίζουν και στόχους και μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων με στόχο την πρόληψη και απάλυνση μετριασμό των επιπτώσεων. Αλλά οι στόχοι αυτοί, καθώς και τα μέτρα, πρέπει να τίθενται με ευθύνη των κρατών μελών και πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες. Από τα έγγραφα που υπευλήθησαν από τις γαλλικές αρχές μέχρι στιγμής, ο ποταμός Όρμπ και η περιοχή, στην οποία αναφέρεται ο αναφέρον, γύρω από το Μπεζιέ, περιλαμβάνεται στο, στο χάρτη για τις περιοχές που κινδυνεύουν από τις γαλλικές αρχές. Σε αυτήν λοιπόν τη φάση, επειδή δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών, δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε σε τι βαθμό τα μελλοντικά αυτά προγράμματα θα λάβουν υπόψη την πληροφόρηση του αναφέροντα και τι προτεραιότητες θα θέσουν οι γαλλικές αρχές και πώς αυτός ο ιδιαίτερος κίνδυνος που έχει να κάνει με αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία θα αντιμετωπίζεται στο σχέδιο. Θέλω να αναφέρω ότι τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης και θα είναι δημόσια έγγραφα μετά την ε, έγκρισή τους. Ο αναφέρον επίσης αναφέρεται σε μέτρα που αφορούν την μορφολογία του ποταμού Όρμπα που μπορεί να έχει να κάνει με τη μεταφορά αποθεμάτων ε, λάσπης. Αυτό το θέμα το αντιμετωπίζει η οδηγία η λεγόμενη για τα ύδατα 62.000 όπου ε, απαιτείται από τα κράτη-μέλη να καθορίσουν πολιτική διαχείρισης για, τα, για, τις, ε, για τις κήτες των ποταμών και πρέπει να περιλαμβάνουν και ένα πρόγραμμα μέτρων που να στοχεύουν στη σωστή διαχείριση των υδάτων των νερών. Ο αναφέρον δεν μας έχει χορηγήσει πληροφόρηση που θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα προγράμματα που προτείνουν οι γαλλικές αρχές δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν το θέμα των υδάτων ή που να καταδεικνύουν ότι αντιστρατεύονται τους στόχους της οδηγίας. Με βάση λοιπόν την πληροφόρηση που μας έχει στείλει ο αναφέρον και λαμβάνοντας υπόψη στη τη φάση εφαρμογής ε, της οδηγίας για τις πλημμύρες δεν βλέπουμε κανένα λόγο να αντιμετωπίσουμε τις ενέργειες των γαλλικών αρχών ως παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα οι συνάδελφοι. Μόνο ο κύριος Μάρτιν έχει δει στο λόγο. Ο κύριος Μαρτά. Ο κύριος Μαρτά λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως Γάλλος, όπως είπε πολύ σωστά και ο αναφέρον, βέβαια δεν είναι μόνο θέμα Δυστυχώ της Γαλλίας είναι ένα θέμα που αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολύ ευρύτερο από τη Γαλλία. Όντω πρέπει να καταδείξουμε τις ε, ευθύνε των μεν και των δε και οι γαλλικές αρχές είναι οι δήμοι. Οι δήμοι είναι αυτοί που εκπονούν το χωροταξικό σχέδιο. Οπότε έχουν και αυτοί ευθύνη. Δεν μπορούν υπό το πρόσχημα των πιέσεων που υφίστανται από τους εργολάβους να δέχονται να χτίζεται όπου να είναι χωρίς να αποτιμούν όλους ε, τους κινδύνους που προκύπτουν. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Κόστ. Οι κίνδυνοι και για τους ανθρώπους, οι οικολογικοί κτλ. είναι σοβαροί. Πρέπει λοιπόν πλήρως να πέσει άπλετο φως στα αίτια, όχι μόνο σε πτώση, στα αίτια των πλημμυρών. Πολύ σωστά το τόνισε ο κύριος ε, Κώστ Τις επιπτώσεις όλοι τις βλέπουμε, δυστυχώς. Αλλά είναι πιστεύω πολύ σημαντικό όλες οι χώρες της Ένωσης να αντιμετωπίσουν πραγματικά τα αίτια των πλημμυρών. Των επανειλημμένων πλημμυρών που έχουν τόσες συνέπειες και στο περιβάλλον και στους πολίτες και εμείς εδώ από τις Βρυξέλλες και το λέω με απόλυτα επίσημο και κατηγορηματικό πρόπο επιτέλους να σταματήσουν ουστ στους εργολάβους και τις ομάδες πίεσης. Επιτέλους οι πολιτικοί που είμαστε, ως πολιτικοί που είμαστε, πρέπει να απαιτήσουμε να μην δικαιολογούνται τα πάντα για λόγους επενδύσεων και ο κύριος Κόστ και τα άλλα θύματα της πλημμύρας έχουν δικαίωμα στην αλήθεια, έχουν δικαίωμα οι πολιτικοί σε κάθε επίπεδο, είτε είναι το γαλλικό κράτο, είτε είναι οι Δήμοι, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν όλα τα μέτρα, ούτω ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον να μειωθεί πολύ ο κίνδυνο. Οπωσδήποτε πρέπει να σταματήσουν αυτέ οι πιέσει. Δεν μπορώ να πω αυτά που θα ήθελα να πω, αν μπορούσα να πω αυτό που θέλω να πω για τους, ε, τις ομάδες θα έλεγα πολύ χειρότερα πράγματα. Και τώρα η κυρία Όκεν. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα συνεχίσω στα Δανέζικα, διότι πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί για άλλη μια φορά να πει ότι αυτό είναι ένα καθαρά εθνικό θέμα. Εδώ όμως ε, υπάρχουν κοινέ πρωτοβουλίε στην Ευρώπη για να παρεμποδιστεί ο κίνδυνος των πλημμυρών και αυτό μας το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι τελικά ε, δρούμε μόνο εκ των υστέρων. Δηλαδή ε, αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία όταν πια είναι πάρα πολύ αργά και δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Πριν από λίγε μόνο ημέρε. ήρθαν σε επαφή μου πολίτες από τη Βουλγαρία, οι οποίοι... από τη Βουλγαρία οι οποίοι ζήτησαν να μιλήσουν στην ε, Επιτροπή Αναφορών για μία αποστολή, επιτόπια αποστολή, η οποία υποτίθεται ασχολείται με την αποψήλωση δασών στη Βουλγαρία. Ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα και το οποίο οδήγησε σε τραγικές πλημμύρες. Εμείς λοιπόν ε, παρεμβήκαμε, τελικά ε, μπορέσαμε κάπως ε, να αποφύγουμε και να παραποδίσουμε την αποψήλωση και δεν προέκυψε αυτή η πλημμύρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δραστηριοποιείται περισσότερο και το θέμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Να μην επανέλθω σε αυτά που ακούσαμε ήδη. Μπορεί να μην συμφωνώ με όλες τις πολιτικές επιλογές ε, του συναδέρφου Μαρτάν, Συμφωνώ με ένα μέρος των όσων είπε. Και θέλω να του πω ότι ξεχνά ένας από τους κύριους λόμπιστ που στρέφεται στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι το γαλλικό κράτος. Όντω, πολλέ φορέ υπέστη πλημμύρε η χώρα μα τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε εβδομάδε και είδαμε στην τηλεόραση τον ένα μετά του άλλου του πολιτικού να ζητούν κατεπηγόντω παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν ή πλημμύρες και κίνδυνοι για πλημμύρες. Οπότε ακόμα και αν δεν είναι άμεση αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή θέτει το πλαίσιο. Οι χώρες μέλη είναι εκείνες οι οποίες θέτουν σε εφαρμογή μέσα σε αυτά τα πλαίσια στρατηγικές πολιτικές για να μην έχουμε κάθε χρόνο τις τραγικές συνέπειες των πλημμυρών με νεκρούς και με, τεράστια, με τεράστιες οικονομικές απώλειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει επιδοτήσεις για να κάνει επενδύσεις για να αποφύγει τις συνέπειες από τις πλημμύρες αυτές. Άρα εμπλέκεται εδώ η Ευρώπη. Και κάτι άλλο όσον αφορά την συγκεκριμένη αναφορά του κύριου Κοστ Ακόμα και αν δεν είμαι ειδικό για την λειτουργία του ποταμού Ορμπο, αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να γράψει στο γαλλικό κράτος για να το υποχρεώσει, αν μη τι άλλο, να απαντήσει στις ερωτήσεις του κύριου Κώστα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο αυτά τα οποία ζητάει είναι έτσι δεν είναι. Δεν είμαι ειδικό, αλλά ένα από τα πιο φοβερά πράγματα για τους συμπολίτε μας και γι' αυτό αναγκάζονται και φτάνουν στη δικιά μας Επιτροπή Αναφορών, εγώ βέβαια μόνο αναπληρωματικός είμαι εδώ, είναι γιατί ακριβώς διαπιστώνουν οι πολίτες ότι τα κράτη τους δεν τους απαντάνε ή του στέλνουν ένα τυπικό γράμμα από το τελευταίο τροχό της αμάξης των υπηρεσιών τους ή δεν απαντούν ποτέ. Αυτή είναι μια μεγάλη απογοήτευση για τους πολίτες. Οπότε αν μη τι άλλο, ο κύριος Κώστα θα πρέπει να πάρει σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτά που λέει στέκουν ή δεν στέκουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε αν αποφασίσουμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή ή και αν δεν την κλείσουμε, η Επιτροπή να ζητήσει από το γαλλικό κράτος να απαντήσει συγκεκριμένα στον κύριο Κώστα. Τουλάχιστον αυτό. Πρόεδρος. Καλώς. Έτσι ολοκληρώνω εδώ τον κατάλογο μιλητών που είχα για αυτό το θέμα. Και στρέφομαι σε εσά κύριε Κώστα. Για να ολοκληρώσουμε την εξέταση της αναφοράς σας. Αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, μπορείτε. Δύο λεπτά το πολύ όμως, ε. Μία πρόταση έχω να πω μόνο, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τα ρεύματα του Ροδανού και του Βαλής και τα λοιπά που μπλοκάρονται. Μέχρι την Αλμερία και το Μαρόκο φτάνουν οι συνέπειες. Αυτό μόνο να σας πω. Το σκάφος ΜΕΝΤ έκανε διάφορες έρευνες και οι εικόνες του πήγαν παντού για τις συνέπειες που έχουν οι καταρακτώδεις βροχές στο Ροδανό και αλλού. Συνεπώς, δεν είναι πρόβλημα της Γαλλίας μόνο, είναι πρόβλημα της Ευρώπης ολόκληρης, για να μην πω ολόκληρης της Μεσογείου. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ήταν μια παρένθεση αυτή που θέλω να κάνω. Je vous remercie, monsieur. Okay, so... Καλώς. Πώς να συνεχίσουμε τώρα από αυτό. Προτείνω το εξή. Προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να στείλουμε επιστολή στις γαλλικές αρχές με την οποία να υπογραμμίζουμε αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Λαβριέ και προκειμένου να διευρεθεί και το εύρος της εξέτασης σύμφωνα με τις επιθυμίες του κύριου Μαρτά. Δηλαδή να ζητήσουμε πέρα από την μελέτη αυτή από το τμήμα ε, πολιτικών που βρίσκεται στην αίθουσα αυτή να γίνει μια μελέτη για τη διαχείριση πλημμυρών. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις πλημμύρες. Έτσι ξεπερνάμε το, τα στενά πλαίσια της γαλλικής περίπτωσης και καλύπτουμε και άλλες χώρες. Αυτό προτείνω εγώ να κάνουμε. Συμφωνείτε ή έχετε να προτείνετε κάτι άλλο. Συμφωνούμε. Καλώς. Ευχαριστώ. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά. Σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη. Αναφορά 1484 του 2008 της κυρίας Κατρίν Λεκόντ σχετικά με τις επιπτώσεις της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην υγεία των κατοίκων που διαμένουν πλησίων του αεροδρομίου Σάρλ Τεκόλ Ροασί. Είναι εδώ η αναφέρουσα σωστά. Πού είναι? Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε λίγο χρόνο για να έρθω και να σας παρουσιάσω την κόλαση που ζω 18 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Σάρλ Ντεγκόλ στο Ρουασί της Γαλλίας. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους που είναι θύματα της σχετική αυτής ρήπανσης έρχονται το ένα μετά το άλλο τα αεροπλάνα πάνω από τα κεφάλια μας. Το 2012 το ύψος ήταν πολύ χαμηλό και μετά από τις τελευταίες εκλογές τον Απρίλιο χαμηλώθηκε ακόμα το ύψος. Ήταν 300 μέτρα δηλαδή το 2012 και βιώθηκε ακόμα περισσότερο. Βέβαια όλα τα θύματα δεν έχουν τη δυνατότητα να πούν, να κάνουν τίποτα. Εγώ εδώ τους εκπροσωπώ. Έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και το δικαίωμα στη ζωή πάνω απ' όλα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Ένα βουλευτή από το Ιβάλντουάζ έλεγε πριν από λίγο ότι είναι οι ελεγκτέ που διαχειρίζονται την ε, κυκλοφορία των αεροπλάνων. Ναι, αλλά ποιο ε, ορίζει τι διαδικασίε. Εγώ ζω στην οικογενειακή κατοικία, είμαι 60 χρονών, Γαλλίδα και αγωνίζομαι εδώ και χρόνια. Γράφω στου πολιτικού, του καλώ να έρθουν επί τόπου κλπ. κλπ. Γιατί θέλω όλη αυτή την ε, ιστορία να μπορώ να την διαχειριστώ και να την καταλάβω καλά. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι όταν χρησιμοποιήθηκε το νότιο τμήμα του αεροδρομίου ο οικισμός υπήρχε ήδη εκεί. Εδώ και 17 χρόνια λοιπόν ενημερώνω για τις συνέπειες αυτής της, ε, αυτών των αεροπορικών ε, διαδρομών που μας οδηγούν να μπορούμε πολύ δύσκολα να ζήσουμε εκεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομείο κλπ. κλπ. Πρέπει να λυθεί υπόψη αυτή η κατάσταση κατεπηγόντω. 400 αεροπλάνα καθημερινά, αν όχι και περισσότερα, τα οποία θορυβούν πάνω από το κεφάλι μου, σαν να έχω καταιγίδα, που με ξυπνάνε τη νύχτα ξαφνικά. Περιμένω κάθε φορά το επόμενο αεροπλάνο σε απελπισία που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Αυτά τα πράγματα τροποποιούν το νευρικό σας σύστημα, τον συναισθηματισμό σας. Μας εμποδίζουν να διαβάζουμε, και μας προκαλούν αλλεργίες και μας αποξενούν και από την οικογένεια που δεν μπορεί να μένει πια σε αυτό το σπίτι. Είχο, έχω αλλεργίες από τα τέλη του 1997 τη νύχτα, η μυρουδιά της κυροζίνης με ενοχλεί. Στο κήπο τα ρούχα που κρεμάω για παράδειγμα που έχω πλύνει έχουν τα ίχνη της κυροζίνης. Όλα αυτά με σκοτώνουν σιγά σιγά, με κάνουν να μισώ τον ήλιο που ανατέλει από την Ανατολή γιατί από εκεί έρχονται οι προσγειώσεις πολύ θα ήθελα να σας βάλω να ακούσετε αυτά που έζησα σήμερα το πρωί στις 4 το πρωί. Αλλά δεν γίνεται. Όπως γνωρίζετε, οι χαμηλές πτήσεις στα 900 μέτρα είναι ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τα αεροπλάνα περνάνε το ένα μετά το άλλο πάνω από το κεφάλι μου. Κάποιοι μπορεί να κάνουν οικονομίες με αυτόν τον τρόπο, αλλά οικονομίες μετράνε περισσότερο από τη ζωή. Δεν είναι πολύ υπεύθυνο αυτό. Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι δεν μπορείτε εσείς να αισθανθείτε και να καταλάβετε αυτό που σας περιγράφω και αυτό που ζω. Μόνο αν έχετε ζήσει κι εσείς μια παρόμοια κατάσταση. Όμως, ό,τι και αν ε, μπορεί να πει ο καθένας για να προστατευτεί από τις οχλήσεις αυτές, πολλές μελέτες έδειξαν ότι τελικά επηρεάζουν τον ίδιο τον εγκέφαλο. Σήμερα κανένας από εμά δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα. Επίσης, η ηχητική αυτή ρήπανση είναι μια συνεχής επίθεση. Όσο για τα χημικά που αναπνέουμε είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλώς κάτι άσχημο που αναπνέουμε. Έχουν γίνει μελέτες για να δούνε ποια είναι η χορύπανση. Μόνο που έγινε εκεί που δεν υπάρχει χειρότερη ηχητική ρήπανση, αλλά σε δημόσιους χώρους. Που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα τελικά δεν είναι ακέραια, δεν είναι αντικειμενικά. Εγώ κοιμόμουν στον πρώτο όροφο της κατοικίας μου. Έχασα τις δυνάμεις μου και την εγκατέλειψα όμως το 2007 και πήγα να κοιμάμαι στο υπόγειο σε ένα μικρό δωμάτιο που απομόνωσα με ένα πολύ μικρό παράθυρο για να αναπνέω που και που τον αέρα, αλλά έναν αέρα που πραγματικά δεν είναι για να αναπνέει κανείς. Όλα αυτά μου κόστησαν 10.000 ευρώ. Βέβαια ο θόρυβος μπαίνει από τη σκεπή, από τον εξαιρισμό, από τα παράθυρα. Πώς είναι δυνατόν να κοφεύουν οι αρχές σε μια τέτοια κατάσταση όπως είναι η δικιά μου και άλλων σαν και εμένα. Οι λύσεις που προτείνουν σε αυτούς που ζουν ακόμα πιο κοντά στην πίστα του αεροδρομίου ποια είναι, είναι να βάλουν ε, ε, δίπλα τζάμια. Μα είναι αυτή η λύση. Ε, η δικιά μου κατοικία βρίσκεται στη ζώνη Δέλτα του Πέμπε που είναι περίεργο που βρίσκεται εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Γαλλία έχει προειδοποιηθεί ότι δεν τηρεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, ηχητική και τη χημική ρήπανση. Η υγεία μου, η οικογένειά μου, το περιβάλλον μου, η περιουσία μου καταστρέφεται. Η ζημιά αυτή 17 χρόνια γίνεται μέρα τη μέρα. Πώς μπορεί κανείς να την υπολογίσει τη ζημιά αυτή. Νομικά μέσα υπάρχουν, αλλά παραβιάζονται από τους πολιτικά υπεύθυνους, από το χαλικό κράτος και από τους συνενόχους τους. Στο άρθρο 24, για παράδειγμα, της ε, Παγκόσμιας Δήλωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έκριναν τα Ηνωμένα Έθνη 1948 που λέει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση ή το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδιών Ελευθεριών που μιλάνε για το σεβασμό της οικογενικής και ιδιωτικής ζωής η οδηγία του Μαρτίου του 2012 που μιλάει για κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να μην γίνεται εκμετάλλευση που οδηγεί σε χορύπανση κτλ. Που δημιουργούνται από την αεροπορική κυκλοφορία και λέει ότι πρέπει όλα αυτά να προστατεύουν την υγεία, ενώ εδώ πρόκειται για την εσωτερική αγορά. Υπάρχει και το άρθρο 1 της Χάρτας για το Περιβάλλον που εγκρίθηκε το 2005 που λέει ότι όλοι πρέπει να ζουν σε ένα περιβάλλον που σέβεται την υγεία. Και το άρθρο L112 του κώδικα για το περιβάλλον που λέει ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και ισορροπημένο ανάμεσα στην Ήπεθρο και τις αστικές περιοχές και ότι όλοι πρέπει να φροντίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος. Και ότι είναι χρέος να φροντίζουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως οι υπεύθυνοι δεν το κάνουν αυτό. Αλλά ευνοούν τις μεταφορές αυτές που ρηπαίνουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις παρά τις διεθνείς ε, δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Γαλλία. Όλα αυτά παραβιάζονται. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να μπορώ να στηριχθώ στη δικιά σας βοήθεια στα διαβήματα που κάνω. Να ξέρετε ότι έτσι καλώς η οικονομία δεν αντικαθιστά τη ζωή και δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνονται σε βάρος της ζωής μας και να θυσιάζεται ο κόσμος ο οποίο πια δεν έχει δικαιώματα στον ύπνο, ούτε στην ανάπαυση, ούτε στην ησυχία, ούτε στον καθαρό αέρα. Ευχαριστώ κυρία μου. Ξέρω ότι έχετε υποφέρει πολύ. Και τώρα λοιπόν στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Δεζέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω λιγάκι για το ηχητικό στοιχείο αυτής της αναφοράς και αν θέλετε μπορεί μετά ο συνάδελφός μου να αναφερθεί περισσότερο στο θέμα της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαφύλαξη ε, της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, κυρίως στην προστασία τους από την ηχορύπανση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις επιζήμιες συνέπειες του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί προβλέπεται σαφής δέσμευση ότι επιθυμούμε να μειωθεί αισθητά η χορύπανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να αναθεωρήσουμε αυτό που έχει διατυπωθεί ως κατευθυντήριες γραμμές για το θόρυβο κατά τη νύχτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί προκύπτουν σαφώς οι ζημιές στην ανθρώπινη υγεία από την ηχορύπανση. Ας πάμε τώρα στην κοινοτική νομοθεσία που ισχύει σε αυτόν τον τομέα. Η αξιολόγηση λοιπόν του θορύβου νομοθετείται από την περίφημη οδηγία του 2000 ε, σχετικά με την ηχορύπανση. Σε αυτή λοιπόν την οδηγία υπάρχουν δύο σαφείς ε, διατάξεις για τα κράτη-μέλη. Πρώτον, ότι πρέπει να χαρτογραφούν την ηχορύπανση, να τη μετρούν και να τη χαρτογραφούν και δεύτερο βήμα με βάση αυτό το στρατηγικό χάρτη καλούνται τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν προγράμματα δράσης για να διαχειρίζονται την ηχορύπανση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι η οδηγία αυτή αφήνει με διακριτική επιχέρεια στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν μόνα τους για τις ανώτατες τιμές από τις οποίες και μετά θα δραστηριοποιούνται. Επίσης, η οδηγία αφήνει διακριτική ευχαίρεια στα κρατημέλη τα μέτρα που θα συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα δράσης που θα εκπονήσουν. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, το Ροϊσί που είναι κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, μέχρι τώρα η Γαλλία πράγματι έχει χαρτογραφήσει την ηχορύπανη στην περιοχή, έχει καταθέσει το σχετικό χαρτί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο, στο ευρύ κοινό ε, και εκεί βλέπουμε ότι πράγματι θα πρέπει να υλοποιηθούν και υλοποιούνται κάποιες προδιαγραφές. Όμως η Γαλλία δεν έχει ε, υποβάλει πρόγραμμα δράσης με βάση αυτό το χάρτη. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μια επιστολή, ε, προειδοποιητική επιστολή στην Πούμε προς τη Γαλλία. Μετά το Φεβρουάριο του 2014 η Γαλλία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόγραμμα δράσης για το αεροδρόμιο υπάρχει αλλά μέχρι τώρα μόνο σε μορφή σχεδίου και αυτή τη στιγμή υπάγεται στη διαδικασία διαβουλεύσεων που προβλέπεται από την οδηγία. Η Επιτροπή λοιπόν θα παρακολουθήσει την κατάσταση, θα περιμένει το τελικό πρόγραμμα δράσης που θα καλύπτει τις ε, ε, προδιαγραφές που προβλέπονται στην οδηγία. Επαναλαμβάνω όμως, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να επηρεάσει ως προς τα μέτρα που θα αποφασίσουν οι γαλλικές αρχές να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα δράσης. Αυτά μέχρι τώρα σχετικά με την οδηγία περί χορύπανσης. Αναφέρουμε σε μια άλλη, στην 30 του 2002 και εκεί προβλέπεται προβλέπονται περιορισμοί με, λόγω της χορύπανσης στα κοινοτικά αεροδρόμια. Αυτή η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν την αποκαλούμενη ισορροπημένη προσέγγιση οποτεδήποτε επιλαμβάνονται του θορύβου στα αεροδρόμια λόγω υπερβολικής κίνησης. Στην πραγματικότητα αυτή η οδηγία σημαίνει ότι στα αεροδρόμια όπου υπάρχει πρόβλημα θορύβου τα κράτη-μέλη δίνανται να λάβουν μία σειρά λειτουργικών περιορισμών που αφορούν και στα θορυβόδια αεροσκάφη, ενώ παράλληλα ε, πρέπει να προσαρμόζονται και σε κάποιες διατάξεις περί κοινής αγοράς. Εδώ λοιπόν προβλέπεται το μέγιστο δυνατό περιβαλλοντικό όφελος με τον πιο προσιτό τρόπο. Οι γαλλικές αρχές έλαβαν τέτοια μέτρα μείωσης ε, του θορύβου λόγω της οδηγίας και η Κομισιόν πρόσφατα αναθεώρησε ε, αυτή την οδηγία που σας προανέφερα, η καινούργια θα εκπονηθεί το 2016. Αυτό ο νέος κανονισμός είναι, γιατί θα είναι κανονισμός, θα ενισχύει το ρόλο των αξιολογήσεων ω προς τη ζημιά στην υγεία και αυτέ οι ζημιές σε σχέση με την ηχορύπανση. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε για το θέμα του θορύβου, αλλά αν θέλετε ο συνάδελφό μου μπορεί να τοποθετηθεί για το θέμα της ποιότητα της ατμόσφαιρας. Πρόεδρος, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παραπέμπω στην γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πολύ ανοιχτή και ξεκάθαρη. Αναφέρει ότι η επιστολή προς τις γαλλικές αρχές δεν ελήφθη υπόψη και η Κομισιόν δεν πήρε κανένα πρόγραμμα δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου. Παρότι θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα δράσης να έχει ήδη υποβληθεί από το 2013. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η γραπτή απάντηση που λάβαμε είναι πολύ ικανοποιητική. Ας καταφύγουμε σε αυτή γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τώρα όμως μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στην άδελφη, παρακαλώ. Ε, θα ήθελα, λέει η κυρία Πιτέρα, να πω το εξής. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να εξαφανιστεί ένα αεροδρόμιο, αυτό είναι ε, μη ρεαλιστικό. Οι τεχνικές ε, προδιαγραφές εξαρτώνται βέβαια από το περιβάλλον. Ξέρετε και στη Βαρσοβία ε, είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε ένα αεροδρόμιο που είναι αρκετά κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτό το αεροδρόμιο πράγματι προκαλούσε πολύ μεγάλο θόρυβο. Σήμερα όμως σε αυτή την περιοχή δεν κατοικεί κανείς πλέον. το κράτος ενίσχυσε τους κατοίκους για να αγοράσουν αλλού κατοικίες. Και οι κάτοικοι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Εγώ έχω μία ερώτηση. Ξέρετε, πράγματι όλοι ξέρουμε ότι μπορούν να υποβληθούν πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Έχω όμως μία ερώτηση προς την αναφέρουσα. Την εξής. Εσείς κάνατε κάτι έναντι των γαλλικών αρχών, στραφήκατε έναντι των αρχών αυτών για να ζητήσετε αποζημίωση, γιατί είναι προφανές ότι η περιουσία που έχει κανείς σε ένα τέτοιο χώρο υποτιμάται, χάνει την αξία της η περιουσία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν εσείς λάβατε μέτρα που είναι απόλυτα φυσιολογικά ε, σε μια προηγμένη χώρα. Ζητήσατε αποζημίωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο ρεαλιστικό να στραφείτε στις γαλλικές αρχές. Και τώρα η κυρία Ντατή, δεν σας βλέπω, αλλά α, βλέπω εκεί είστε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι όλα υπόθηκαν, ιδιαίτερα από την κυρία Λεκόντ. Βεβαίως η ποιότητα του αέρα είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Παρισίων και καταλαβαίνω την οργή που εκφράζει η αναφέρουσα και ως ε, Ευρωβουλευτής της περιοχής αυτής. Όλες αυτές οι οχλήσεις οπωσδήποτε έχουν τραγικές και ουσιώδες επιπτώσεις στην υγεία. Οι κάτοικοι της περιοχής επίσης ε, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για την ποιότητα του αέρα. Αυτό είναι κάτι που μας ε, αφορά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά οι οχλήσεις για αυτούς που είναι πολύ κοντά στο Ρουασί Σαλντογκόλ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητα του αέρα, έχουν να κάνουν και με την ήχορύπανση. Η επίπτωση των δραστηριοτήτων του αεροδρομίου στην ποιότητα του αέρα είναι αισθητή ακόμη και 5 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο. Και γύρω από την πλατφόρμα του αεροδρομίου έχουμε 118 δήμους και γύρω στο 1,8 εκατομμύρια κατοίκους. Η πλατφόρμα Γουασί Ουασί-Σόντεκολ είναι ιδιαίτερα ρηπαντική και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όχι μόνο τις πρωτοβουλίες και όλες τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτή τη κυρίας Λοκόντα προσπαθώντα να μειωθεί η ατμοσφαιρική μόνηση και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Καταλαβαίνω πολύ καλά λοιπόν την, την ε, πρωτοβουλία αυτή και ο, η χορύπανση είναι και αυτή η ρήπανση. Είναι ουσιώδης και πραγματική. Η χορύπανση είναι θέμα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, πάνω από 44% των περίοικων δηλώνουν ότι θα ήθελαν να μετακομίσουν. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ο θόρυβο από τα αεροπλάνα είναι ο πρώτο λόγο που αναφέρουν για να εξηγήσουν αυτή του την απόφαση. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την οποία ψηφίσαμε για το καλό των συμπολιτών μα. Δεν είναι απλώ υποχρέω... καθήκον, είναι υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει Επειδή ε, έχουμε καθυστερήσει πολύ και επειδή η κυρία Λεκόντ, η αναφέρουσα, ήδη μίλησε αρκετά, ίσως θα μπορούσαμε να κλείσουμε την εξέταση της ε, αναφοράς αυτής και αυτό που άκουσα από την Επιτροπή σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή μέχρι οι γαλλικές αρχές να μας υποβάλουν επιτέλους την αντίδρασή τους ε, σε αυτήν την κλίση προς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως μας υποσχέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη αλλά δεν έχουν ακόμη λάβει το συνοπτικό πρόγραμμα. Ήδη το Φεβρουάριο απάντησαν σε εμά, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν υποβάλει αυτό το πρόγραμμα. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Νοέμβριο είναι πολύ ο χρόνο. Προτείνω λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, υπό εξέταση, και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει αυτό το συνοπτικό πρόγραμμα δράσης από τις Γαλλικές Αρχές, εμείς ως Επιτροπή Αναφορών, θα θέλαμε ιδιαίτερω να το εξετάσουμε κι εμείς και θα μπορούσαμε και εμείς βεβαίως να αποστείλουμε μια επιστολή στις ε, Γαλλικές Αρχές για να τους μιλήσουμε για την ανησυχία μας για το επίπεδο ηχορύπανση και γενικά ρήπανση. Εντάξει, συμφωνείτε? Υποθέτω ότι η σιωπή είναι συνένεση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Για να φέρουσα, Παρακαλώ. Άκουσα ότι μου ζητήθηκε αν είχα εξετάσει και άλλα διαβήματα. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει μήνυση στη Γαλλία. Πρόεδρος, μα είμαι πεπισμένο ότι θα κάνατε οπωσδήποτε ό,τι μπορούσατε να κάνετε. Ναι, αλλά πώς θα με αποζημιώσουν για τα 17 χρόνια και τα υπόλοιπα όσα μου μένουν, γιατί δεν είμαι πλέον νέα πώς θα ε, επιτύχω. Ευχαριστώ. Καταλήγουμε με την ε, εξέταση του θέματος αυτού και περνάμε στο επόμενο θέμα. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση, διότι από κοινού πρέπει όλοι να το επιχειρήσουμε. Μαζί με την Κομισιόν και τι Γαλλικές Αρχές. ευχαριστώ πολύ. Και τώρα λοιπόν να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. Αναφορά 1707 της κυρίας Ζαμπίνε Κούριο Μακνίου που ζητάει να καταργηθεί η υιοθεσία χωρίς γονική συνένεση και την αναφορά 2468 κάθος 13 του Roy Fox, Βρετανικής Θαγένειας, σχετικά με τις καταναγκαστικές υιοθεσίε του Ηνωμένου Βασίλειο. Νομίζω ότι είναι παρόντες οι αναφέροντες. Α, μάλιστα, καλώ ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο σε εσά απευθείας. Λάβαμε μια επιστολή από τον Υπουργό Ιούλιος 14. Έχει διανεμηθεί. Μόλις τώρα τη λάβαμε εμείς, οπότε τώρα μόλις διανεμήθηκε την έχετε στο έδρανό σας. Να δώσω το λόγο, να δώσω συγγνώμη το λόγο, στη κυρία Ζαμπίνε Κούριο Μακνίου. Καλησπέρα. Λέγομαι Ζαμπίνε. Γερμανικό όνομα. Κούριο είναι σλαβικό. Αυτό εξηγεί το πάθος μου. Και ήμουν παντρεμένη με έναν Σκοτσέζο. Αλλά παρόλα αυτά διατήρησα την γερμανική μου υπηκότητα. Είμαι εδώ από πλευρά τη Ένωση των Φίλων των Μακέντζη, την οποία ίδρυσα και έχουμε και ένα ιστοχώρο. Είμαστε νομικοί σύμβουλοι κυρίω που βοηθάμε τα θύματα ιδιαίτερα των οικογενειακών δικαστηρίων, σε κάθε επίπεδο. Εμείς ιδιαίτερα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, δεν, γενικά δεν συμμετέχουμε τόσο πολύ σε υποθέσεις επιμέλειας μεμονωμένες, αλλά έχουμε υποβάλει μια μελέτη όπου περιγράφουμε ότι υπάρχει συστηματική ε, διαδικασία για την αρπαγή παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έκτοτε ε, έγιναν ορισμένα πράγματα, ιδιαίτερα στη διεθνή ε, σύσκεψη για ε, την αφαίρεση παιδιών στην Πράγα. Η Επιτροπή Μαρτίου συστήθηκε από 30 γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους και που είχαν μεγάλες προσδοκίες από την δική μου αναφορά. Δεν υποβάλαμε λοιπόν μόνο μία έκθεση, αλλά και ένα φάκελο 12 ε, σελίδων με στοιχεία και υποβάλαμε και ένα αριθμό υπογραφών. Και το σύνολο των 4 ή 5 αναφορών είχαν συλλέξει πάνω από 8.000 υπογραφές. Η προηγούμενη επιτροπή μας είχε υποσχεθεί μία ε, αποστολή εξέβρεση στοιχείων. Περιμένουμε ακόμη. Τα έξι λεπτά της έντονης παρουσίασής μου ε, τα ε, έγραψαν διάφορες τηλεοπτικές κάμερες και παίχτηκαν, αλλά η Επιτροπή μου είπε ότι δεν μπορεί να δώσει συνέχεια. Έλαβε μια επιστολή που το έλεγε. Παράλληλα, μίλησα και σε Πορτογάλους γονείς που τους είχαν αφαιρεθεί τα πέντε παιδιά τους και οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία της κομιτείας του Lincoln, Lincolnshire γιατί ανήκαν στην ε, ομάδα για την καταπολέμηση των καταναγκαστικών υιοθεσιών και βλέπουμε ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζονται ως εγκληματίε. και τα παιδιά. Τα νεότερα παιδιά υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί τον, ε, στις 17, συγγνώμη, τον Οκτώβριο του 17 ένας ε, διπλωμάτης από την Πρεσβεία συναντήθηκαν με την αστυνομία του Λίνκον και ε, τους υποσχέθηκαν ότι τα παιδιά θα επιστραφούν σε ένα πορτογαλικό ίδρυμα, αλλά αυτό ακόμη δεν έχει συμβεί. Ωστόσο, ο πατέρας έκτοτε απολύθηκε δύο φορές, διότι οι κοινωνικοί λειτουργοί της περιοχής τηλεφώνησαν στους εργοδότες και, του είπαν, και τους είπαν να απολυθεί. Ένας ουαλός πατέρας που ήταν παρόν μαζί μας και απεγνωσμένα ήθελε να δει τα παιδιά του και αυτός τιμωρήθηκε επειδή ήρθε εδώ στις Βρυξέλλες γιατί και δεν του επιτράπηκε να επισκεφθεί το γιο του στην, στα γενέθλια του γιού του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Αυτή η απόπειρα αυτοκτονία δεν είναι η μόνη. Σε αυτή την περιοχή της Ουαλίας, στο Καρνάβονσια, έχουν γίνει και άλλες τέτοιες απόπειρες αυτοκτονίας. Οι φίλοι μου από την οργάνωση Μακένζη, που ήρθαν μαζί μου στις Βρυξέλλες, διαπίστωσαν κατόπιν ότι έγιναν και άλλες δύο δολοφονίες, ε, συγγνώμη, ε, αυτοκτονίες μεταξύ των ε, συμμετεχόντων σε αυτήν την, ε, σε αυτή την ομάδα. Και ε, άλλες ποινές έχουν επιβληθεί στους Βρετανούς υπηκόους που έρχονται στις Βρυξέλλες να διαμαρτυρηθούν. Και μας προτείνεται να ασχοληθούμε κυρίως με τα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Το γεγονός λοιπόν ότι παιδιά από άλλες χώρες δίδονται για υιοθεσία σε Βρετανούς γονείς και σημαίνει αυτό ότι εκτίθενται σε άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία ενδεχομένω, άλλες συνήθειες. Αυτό αναφέρθηκε σε αυτή τη διάσκεψη στην Πράγα. Εκεί μια κυρία από τη Σλοβακία ενεπλάκη σε αυτήν την ε, περίφημη υπόθεση όπου δύο παιδιά επεστράφησαν μετά την καταναγκαστική υιοθεσία μετά από 920 μέρες που τα είχαν αναλάβει οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ο Τζον Χέμινγκ επίσης έχει τα στοιχεία για αυτά που έχουν συμβεί σε 100 οικογένειες στην Ιρλανδία. Ίσως να έχετε ακούσει και για την υπόθεση Άσια King που, ήταν, ε, που είναι αυτό το παιδί που έχει καρκίνο και του οποίου οι γονείς φυλακίστηκαν. Έχουμε λοιπόν ε, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να ε, βρει μητέρες οι οποίες έχουν φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες χώρες αλλά οι μητέρες και οι γονείς που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους. Η διάσκεψη του, της Πράγας αναφέρθηκε επίσης και στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2012 και που σχετίζεται και με τη συμβάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των παιδιών. Αν έρθετε στο Λονδίνο, μπορεί να έχετε πάρει τον υπόγειο. Πολλέ φορέ εκεί στον υπόγειο λέει προσοχή στο κενό ανάμεσα στην πλατφόρμα και το τρένο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κενό που πρέπει να προσέχετε. Είναι το κενό ανάμεσα στον νόμο και την πραγματικότητα. Πώ εφαρμόζεται ο νόμο. Αυτό το κενό είναι τεράστιο. Και ελπίζω ειλικρινά η Επιτροπή να σημειώσει αυτά που λέω, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αρκετά σε επαφή με τα θύματα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που η Επιτροπή Αναφορών είναι εδώ και ακούει τα θύματα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Η Νάταλη Στόκουελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω την κυρία Κούργιο Μακνίλ για την ε, εμπεριστατωμένη παρουσίαση που μας έκανε, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά τα θέματα ήδη συζητήθηκαν ε, στις συνεδρίες του Μαρτίου της Επιτροπής Αναφορών και πιστέψτε με, απασχολούν την Επιτροπή. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά λαμβάνοντα σε υπόψη ένα πράγμα κατά κύριο λόγο, των συμφέρων του παιδιού. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου στις συνεδρίες του Μαρτίου. Τα έχουμε πει εξάλλου και σε ανταλλαγή ε, επιστολών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους συναδέλφους. Ούτε θα επαναλάβω την επίσημη απάντηση που σας δόθηκε γιατί φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να τα ξανακούσετε όλα αυτά και πιστέψτε με ήταν και για μένα πάρα πολύ επώδυνο να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Λόγω της σοβαρότητας ε, του θέματος είτε είμαστε αρμόδιοι είτε όχι ήρθαμε σε επαφή με τις Βρετανικές Αρχές το ίδιο έπραξε και η Επιτροπή Αναφορών. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και εδώ αναφέρομαι στην επιστολή που ανέφερε και η Πρόεδρος που διανεμήθηκε και σήμερα αναφέρει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αυτός είναι ο πρωταρχικός ε, παράγων και παραθέτω οι οικογένειες ε, θα πρέπει να λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για να διαφυλάστε το συμφέρον του παιδιού και τέλος της παράθεσης. Καταλαβαίνω, είπατε ότι αυτό δεν συμβαίνει, αυτή την εμπειρία έχετε κάνει και να σας πω λοιπόν προσφέρω να συναντηθούμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε βάθος. Οι συνάδελφοί μου, οι αρμόδιοι θέματα δικαιωμάτων παιδιών θα είναι παρόντες, να τα συζητήσουμε και εν ώψη των κατευθυντήριων γραμμών που προτιθέμεθα να εκπονήσουμε για συστήματα προστασίας. Θα σας ενημερώσω. Σε αυτή τη συνάντηση έχουμε προσκαλέσει και συναδέλφους από την ε, Διεύθυνση 2α ε, σας λέω λοιπόν ότι εκεί σε αυτή τη συνάντηση θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εμπεριστατωμένα πλέον όλα αυτά τα θέματα. Και εμεί ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ε, μπορούν να υποβάλουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Κυρία Σακοράφα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, όταν προσεγγίζουμε ζητήματα που αφορούν σε παιδιά και με αφορμή το συγκεκριμένο, και ειδικότερο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίζω να ξεκινάμε από μια κυρίαρχη και αδιαπραγμάτευτη και διαφημισβήτητη άποψη παγκοσμίω, ότι δηλαδή δεν υπάρχει πιο ιερή σχέση από αυτή μεταξύ του γονιού και των παιδιών. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για να υποστηρίξω όσα λέω, ακριβώ γιατί οι περισσότεροι από εμά σε αυτή την αίθουσα είμαστε γονεί. Απλά θα ήθελα να αναφερθώ σε πρόνοιες που έχουν ληφθεί έτσι ώστε αυτή η σχέση να υποστηρίζεται με κάθε τρόπο άμεσα, ακόμα και όταν οι αντικειμενικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν και δεν το βοηθούν. Αναφέρουμε στις προσπάθειες που γίνονται έτσι ώστε αυτή η σχέση να διατηρείται, ακόμα και σε περιπτώσεις που οι γονείς είναι φυλακισμένοι για βαριά δικήματα που δεν έχουν όμως να κάνουν με, με οικογενειακές παραβάσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι σωστά πράττουμε πάνω σε αυτό και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση η υποβοήθηση του γονιού έτσι ώστε να μπορεί να υπηρετεί το ρόλο του σε περιπτώσεις όπου έχει απομακρυνθεί από αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η ιδιαίτερη σχέση πρέπει να είναι οδηγός και για το πώς προσεγγίζουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνουμε στην προσπάθεια και την αγωνία μας να προστατεύσουμε την τρυφερή ηλικία των παιδιών. Από αυτή την οπτική εκτιμώ ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να τύχει ιδιαίτερη επιμέλεια και από την Επιτροπή μα και να εξεταστεί σε βάθο και μάλιστα όχι μόνο στα στενά νομικά πλαίσια. Ε, δεν θα ήθελα να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα από την πρώτη ανάγνωση αυτού του θέματος και γι' αυτό παρακαλώ για μια πιο ευρία διερεύνηση του θέματος, μιας και έχει προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσον αφορά το εθνικό δίκαιο, πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν στι οικογενειακέ σχέσει. Πρέπει λοιπόν, πιστεύω κυρία Πρόεδρε, να, να εξαντλήσουμε όλα τα εργαλεία και τα μέσα που μας δίνει αυτή η Επιτροπή και αυτό μπορεί να είναι η πρόκληση κανονισμού, οδηγιών για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη ε, και τη σχετική παράγραφο στην απάντηση της Επιτροπής, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ την τελευταία παράγραφο πριν από τα συμπεράσματα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι ενδιαφερόμενοι γονείς ε, που πιστεύουν ότι οι περιπτώσεις υιοθεσία που γίναν χωρίς τη δική του συγκατάθεση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχοντας και λαμβάνοντας υπόψη και το οικονομικό πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι γιατί είναι μετανάστες, να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας οδηγός για μας ε, και να προσέξουμε και να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την υπόθεση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή με την ανοχή τη και τη δική σα, κυρία Πρόεδρε, να μου δίνετε τη δυνατότητα, επειδή πρέπει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να φύγω, να αναφερθώ και σε μια μεθεπόμενη υπόθεση, την υπόθεση 1156 του κυρίου Γιαννόπουλου που παρότι έχω διαβάσει όλο το σχετικό φάκελο και έχω διαβάσει και την αναφορά που έχει γίνει και από το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και από την, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου θα ήθελα να πω ότι για λόγους ευαισθησίας γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει σε χώρες που δεν καλύπτονται από τις δικές της ε, οδηγίες και νόρμες. Αλλά θα έλεγα ότι για λόγους ευαισθησίας απέναντι και στο παιδί αλλά και στην αγωνία του πατέρα θα παρακαλούσα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση για να ξανασυζητήσουμε και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ενεργειών που υπάρχει επαφή μεταξύ του παιδιού και των δύο γονιών, θα έλεγα εγώ, ώστε να εξασφαλίσουμε την απαρκή σχέση του παιδιού και με τους δύο γονείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά Γιαννόπουλου είναι πιο κάτω στην ημερήσια διάταξη. Θα συζητήσουμε αυτά αργότερα, αυτές τις δυσκολίες. Η κυρία Κέρτον Τάλινγκ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε την πρώτη απόφαση που πήραμε σήμερα το πρωί για το ότι οι αναφορές που έχουν να κάνουν με παιδιά πρέπει να προωθούνται, να μπαίνουν πιο πριν στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είπαμε το πρωί. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική απόφαση αυτή που πήραμε. Επίσης, πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα όσον αφορά το Ενωμένο Βασίλειο. Η ανησυχία για το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να κάνει και με ιστορικά γεγονότα, με διασμούς και κακοποίησεις που γινόντουσαν σε διάφορα ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο από παλύτερα και έγιναν και διάφορες έρευνες και εξεταστικές ε, επιτροπές έλαβαν χώρα για τέτοιου είδους καταγγελίες. είναι ένα συναισθηματικά φορτισμένο θέμα αυτό και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις για προβλήματα που δημιουργούνται από τέτοιου είδους υιοθεσίε πρέπει να τα πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Τα δικαιώματα των παιδιών σημαίνει ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού και βάσει αυτού πρέπει να κινηθούμε. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε στις προηγούμενες ανησυχίες της Επιτροπής μας και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Βλέπει κάποια νομική προσέγγιση στο θέμα. Πάντως ο αριθμός των αφορών δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Και συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή που είπε, με την κυρία Σακοράφα, που είπε ότι πρέπει να το δούμε ευρύτερα αυτό το θέμα, όχι μόνο δηλαδή στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά γενικότερα ευρωπαϊκά. Το θέμα δηλαδή της προστασίας των παιδιών, των υιοθεσιών κλπ. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημειώνω αυτό που είπε, ότι είναι δηλαδή εθνική αρμοδιότητα ως επιτοπλίστων. Ναι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ερευνηθεί λεπτομερέστερα το τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους. Είναι ανεβαίσθητο θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με πολύ λεπτό τρόπο, προσεκτικά. Και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να δώσει μια πιο λεπτομερή απάντηση όσον αφορά τις διάφορες περιπτώσεις. Αυτό βέβαια συνδυάζεται και με τις έρευνες που γίνονται για διάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών εκεί. Αυτό είναι το πρώτο μου σημείο. Το δεύτερο θα είμαι πιο σύντομη τώρα κύριε Πρόεδρε. Είναι το ότι προφανώς τίθεται θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας κάθε φορά που έχουμε διασυνοριακές περιπτώσεις. Και πρέπει να έχουμε μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις υιοθεσιών. Μια άλλη μου σύσταση είναι να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την ε, Νομική Επιτροπή για το κατά πόσο πρέπει να ασχοληθούμε το θέμα της διασυνοριακής προστασίας και διασυνοριακών υιοθεσιών στα πλαίσια του Βρυξέλλες 2 αν συνάδει με τον κανονισμό αυτόν δηλαδή που αναθεωρήθηκε. Καλό θα ήταν να περιμένουμε να έχουμε και την απάντηση αυτή, αυτή τη γνωμοδότηση δηλαδή. Ωραία. Παρακαλώ εσείς. Κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ ότι... Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που ακούω εγώ τέτοια πράγματα να συμβαίνουν το 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν άκουσα για τέτοιες ε, υιοθεσίε. Εγώ σκέφτηκα την εποχή του Πινοσέτ στην Αργεντινή, στη Χιλή, όπου χιλιάδε παιδιά μετά την ε, εξαφάνιση των γονιών τους υιοθετήθηκαν. Αλλά ναι, παρόλο που είναι βέβαια πολύ λεπτό το θέμα για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλα αυτά πρέπει να ερευνηθεί ώστε πολύ προσεκτικά και με σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις αυτές. Ομολογώ επίσης ότι προσωπικά πάντα είχα πρόβλημα με την έννοια αυτή ποιο είναι το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, γιατί είναι υποκειμενικό. Εξαρτάται ποιος αποφασίζει ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Δεν ξέρω, ένα κριτήριο είναι να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του παιδιού. Έχω όμως δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί θέλω να καταλάβω καλύτερα. Όταν μιλάμε για αθεσία, μιλάμε για την κλασική υιοθεσία ή μιλάμε για την τοποθέτηση των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και δεύτερον, η υιοθεσία αυτή καθεαυτή, όχι η ανάδοχη οικογένεια, η υιοθεσία δεν απαιτεί μία δικαστική απόφαση και την σύμφωνη γνώμη των γονιών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, μα ακριβώς αυτά γίνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονιών. Περί αυτού πρόκειται. Κοιτάξτε λίγο το σημείο 14 στο φάκελό σας. Θα δείτε, εκεί υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Μια που δεν έχουμε πολύ χρόνο, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στην Γιάννα Τούρνο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τους προελίσσαντες και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πριν από σάντησή μας ε, επικοινώνησα ε, με έναν αρμόδιο στην Αγγλία και μου είπε ότι πράγματι ισχύουν όλα αυτά για την απομάκρυνση των παιδιών. Οι μισές περιπτώσεις ε, εξ αυτών είναι όπως περιγράφονται. Και μια παρατήρηση, ορισμένες υποθέσεις δεν αναφέρονται στην πρεσβεία μας γιατί δεν είναι νόμιμοι οι μετανάστες εμείς ε, οι Εστονοί έχουμε περισσότερα προβλήματα ας πούμε στη Νορβηγία που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Φινλανδία. Η Εστονία έχει περισμένο αριθμό ε, κατοίκων Παρ' όλα αυτά εμείς μπορούμε να αναφέρουμε τουλάχιστον 12 περίπλοκες περιπτώσεις. Υποθέτουμε βέβαια ότι η αριθμή αυτή είναι πολύ ψηλότερη ε, για τις μεγαλύτερες ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες γιατί, για τι ακριβώς διαδραματίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών. Δεν είμαστε σίγουροι για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εκείνοι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι ασκούν το, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Ίσως ε, λοιπόν θα μπορούσαμε να αναθέσουμε μια ειδική μελέτη για αυτά τα θέματα. Και κάτι άλλο ακόμα. Ε, θα ήταν κατά των βασικών ευρωπαϊκών αρχών αν οι άνθρωποι φοβούνταν να επισκεφθούν κράτη όπου δεν είναι σαφής η προστασία των παιδιών. Έχω την αίσθηση ότι οι τοπικές αρχές ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ποικιλομορφία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υπάρχει καλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να είναι πιο σαφείς οι κανόνες για να μην παραβιάζονται και τα δικαιώματα των παιδιών και των γονέων. Με πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Η κυρία Σντανόκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ε, που υποστηρίζουν την αναφορά. Συμφωνώ με τη Σαμπίνε Μακνίλ η οποία έκανε την ανακεφαλαίωση και μας έδωσε πολλές και πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το κεφάλαιο 3 ε, στην παρέμβασή της το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει από τα 28 κρατημέλη σχετικά με την καταναγκαστική υιοθεσία. Υπάρχει η περίπτωση η Μαρτίου, ε, πολίτη από τη Λετωνία που εξακολουθεί να είναι ανοιχτή, να κρεμεί. Σήμερα η Λάλα είναι και αυτή παρούσα. Και αυτό αποδεικνύει ότι δυστυχώς ε, ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά οποτεδήποτε πρόκειται για επικοινωνία με βρετανικές αρχές και πρόθεση μιας αναφοράς. Έχουμε αυτή την επιστολή από τις ε, Βρετανικές Αρχές της 10ης Οκτωβρίου του 2014. Την έχουμε αυτή την επιστολή και δίδεται μία απάντηση στην επιστολή της κυρίας Μασόνη της πρώην Προέδρου της Επιτροπής μας η οποία έστειλε μια επιστολή τον Ιούλιο του 2014. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι δεν γίνονται σεβαστές οι απόψεις της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ε, το πιστεύω αυτό. Αλλά το αρνούνται οι αρχές ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρόλα αυτά, αυτό που παίζει ρόλο στην απάντηση που μας δίδουν είναι ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει απάντηση επί της ουσίας, γιατί αναφέρουν έτσι γενικά ότι πρέπει να αποκτήσουμε την άδεια του ε, δικαστηρίου για να μπορέσουμε και εμείς να προβούμε σε δικές μας έρευνες και να ε, ανταποκριθούμε στην αναφέρουσα. Άρα δηλαδή τι σημαίνουν αυτά. Σημαίνουν ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει έτσι μια πολύ μεγάλη διομορφία. Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και τιμωρίας ε, των, ε, του αναφέροντος ή της αναφέρουσας. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση της λετονής που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα σταματήσω εδώ, πρέπει όμως να σας πω ότι είμαι ευγνώμων απέναντι στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δήλεσε ότι δεν θα αναφερθεί και πάλι στο άρθρο 51 όπου ακούμε ότι η Κομισιόν ασχολείται με θέματα παραβίασης ε, του Οικουμενικού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει μία απάντηση του κυρίου Τίμεμανς που λέει ότι με μεγάλη του χαρά να συζητήσει με την πρόεδρο Επιτροπής Αναφορών κατά το κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα με το άρθρο 51. Ελπίζω λοιπόν, αγαπητή πρόεδρε, να το δείτε το θέμα, να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την αντίφαση που υπάρχει. Πάντως, κατά τη δική μου άποψη, ότι αν έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις από πολίτες ε, ευρωπαϊκών κρατών που ε, διαβιούν στη Μεγάλη Βρετανία, αν υπάρχουν τέτοιου παραβιάσεις, κατ' ουσίαν παραβιάζουν την αρχή ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι παγιωμένη και κατοχυρωμένη αρχή στις ιδρυτικές συνθήκες. Τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ο κύριος Πιταγιά και μετά αν θέλετε κλείνουμε τον κατάλογο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Όλοι έχουν υποθεί, αλλά πρέπει να διαπιστώσω ότι η κατάσταση ελάχιστα είναι ικανοποιητική. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε αυτά. Και κατά την προηγούμενη θητεία τα είχαμε συζητήσει, ότι δεν συμφωνούμε, ότι παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωπαϊκά δικαιώματα, η ευημερία των παιδιών, αλλά δεν έχουμε επιτύχει τίποτα. Στην ουσία είναι ένας φαύλος κύκλος, διότι η Αγγλία κατεβάζει τα ρολά και λέει δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας αφορά αγαπητή Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας θέμα. Και είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το θέμα. Έτσι αντιμετωπίζουν οι αρχές. Ε, οι αρχές λένε μια χαρά είναι τα πράγματα, οι Βρετανικές αρχές. Οπότε θα πρότεινα, Πρόεδρε, να το δούμε πιο κοντά, από πιο κοντά το θέμα αυτό, να κάνουμε μια κρόαση για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχει ανάγκη, πιστεύω, να νομοθετήσουμε από αυτού, αλλά δεν είμαι εμπειρογνώμων. Αλλά κοιτάξτε, η πολιτική, όπως λέμε, ξεκινάει από μια εξέταση της πραγματικότητας. Αυτό το κάναμε. Και αν δεν μας ικανοποιεί η πραγματικότητα, τότε πρέπει να την αλλάξουμε. Το θέμα είναι πώς θα την αλλάξουμε. Και γι' αυτό προτείνω μία ακρόαση. Από κοινού με τους εμπειρογνώμονές μας από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, γιατί είναι πολύ περιπλοκό το θέμα αυτό και πρέπει να θεωρήσουμε ότι ό,τι και να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε, θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε. Ό,τι και να κάνουμε θα υπάρχει ο αντίλογος τα κράτη-μέλη δεν θα συμφωνήσουν και θα καλυφθούν πίσω από τους νόμους τους. Πρέπει να διαπιστώσουμε επίσης ότι τα προβλήματα για τα δικαιώματα των παιδιών δεν αφορούν μόνο τον Ενωμένο Βασίλειο και με την Γερμανία είχαμε προβλήματα και αναφορές και με τη Δανία και πάλι τα ίδια μας λένε και άλλες χώρες. Όχι, είναι δικό μας θέμα, αγαπητή Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε φτάνει η Επιτροπή μας στα όρια των δυνατοτήτων της. Γι' αυτό η πρότασή μου λοιπόν επαναλαμβάνω να κάνουμε μία ακρόαση. Γιατί το πρόβλημα αυτό πιστεύω ότι αξίζει μία ακρόαση, αλλά όχι μόνο μεταξύ μας και με τους συναδέλφους της Νομικής Επιτροπής οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Γιατί πραγματικά είναι πολύ λυπηρό το θέμα αυτό. Μας πονάει οι αναφέροντες να έρχονται και να μας ξαναλένε ωραία, ωραία. Μας εμψυχώσατε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά στην ουσία δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Αυτό με ενοχλεί, με ενοχλεί τρομερά. Κοιτάξτε συνάδελφοι, είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι για τα παιδιά, το μέλλον τους, είναι για τη ζωή και τα δεινά των ανθρώπων. Είναι ένα από τα πιο λεπτά θέματα που μας έχει απασχολήσει ποτέ σε αυτήν την Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε προσεκτικά, με ψυχρό κεφάλι και ε, ζεστή καρδιά. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τον ε, αναφέροντα κύριο Εζίν Λουκανιέγκο Ζωηφέρτης και την κυρία Μπογκουσλάβα Γκλαζένσκα παρούσα και εκείνη, και την κυρία Άστα Ιγναταβίτσε. Παρούσα επίσης βεβαίως. Ωραία. Από πλευράς εκπροσωπώντας την αδελφή σας. Ωραία. Ωραία και θα έχουμε και ένα κείμενο μέσω βίντεο. Ο κύριος Λουκιανέγκο Ζωηφέρτης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην Επιτροπή σας που μου δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά. Είμαι Ολλανδός πολίτης, αλλά ρωσικής καταγωγής και εβραϊκής θρησκείας. Θέλω να αφαιρθώ σε αυτά που υπόθηκαν για την προστασία των παιδιών και για την αντίδραση των ε, Βρετανικών αρχών. Έχω μπροστά μου μία δικαστική απόφαση που λέει πληροφορήσατε τις αρχές, το δικαστήριο, όπου ότι θέλετε να πάτε στις Βρυξέλλες για να μιλήσετε στην Επιτροπή Αναφορών. Σας απαγορεύεται να, να ενημερώσετε για οποιαδήποτε στοιχεία αυτής της υπόθεσης και απαγορεύεται να γνωστοποιήσετε καμία πληροφόρηση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκφράσεις άποψης του γιού μου για, τους, ε, για την υπόθεση αυτή και για όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή και με τους θετούς γονείς, τους παρέθετους γονείς με τους οποίους ε, είχε να κάνει. Μίλησα με ένα νομικό σύμβουλο και μου έδωσε μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση. Αν αναφέρω οτιδήποτε, ο γιος μου μπορεί να εξαφανιστεί. Αν αναφέρω ε, την, ε, τις τοπικές αρχές που εμπλέκονται οι τοπικές αρχές όμως αυτές είναι εκεί. Αναφέρονται στην αναφορά. Αυτή η δικαστική απόφαση δεν έχει ημερομηνία. Και μία άλλη έχει προ έχει λάβει πρώτερη ημερομηνία, είναι προχρονολογημένη 16 Οκτωβρίου. Α, όλα αυτά σημαίνουν ότι η απόφαση αυτή ήταν ήδη έτοιμη πριν την ε, εγκρίνει τυπικά ο δικαστής. Δεν μπορώ να αναφέρω για ποια τοπική αρχή πρόκειται το φοβάμαι για το παιδί μου. 100 και 150 περίπου, έως 150 παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στο Κέντ. Φοβάμαι λοιπόν για το παιδί μου και σας δω συγγνώμη. Έχω ε, όμως ακούσει όμως ότι υπάρχει ένα βίντεο με το παιδί μου και αν πάθει τίποτα το παιδί μου θα σας αποσταλεί το βίντεο αυτό. Κοιτάξτε. Υποχρέωσαν το παιδί μου να πάει σε θετούς γονείς. Χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Ήταν πολύ καλός μαθής ιδιωτικό σχολείο. Ήταν 9 ετών και 7 μηνών. Ο γιος μου, ε, το παιδί μου το ανέλαβαν ε, κάποιες, ε, κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί και εγώ συνελήφθη Είχαν πει ότι δύο παιδιά είχαν κάνει κάποιο αδίκημα κατά της περιουσίας αλλά το άλλο παιδί δεν συνελήφθη. Μία κοινωνική λειτουργός είδε το παιδί μου για 30 λεπτά δύο φορές και λέει ότι εγώ του επέβαλα τη θρησκεία μου γιατί είναι μέλος μιας συναγωγή όπου πηγαίνω και εγώ και εκείνο. Πώς είναι τα συμφέροντα του παιδιού λοιπόν το πρωταρχικό. Δεν μας επιτρέπουν να μιλήσουμε ρωσικά, που είναι η γλώσσα προέλευση. Το παιδί μου είναι δίγλωσο. Διότι η κοινωνική λειτουργία λένε ότι του επιβάλλω τη γλώσσα μου. Μα αφού το παιδί αυτό από τότε που είναι μαζί μου μιλάει τη γλώσσα μου. Που είναι και γλώσσα του. Είναι θέμα διάκρισης λόγος που πρέπει να λόγος που θέλουν να αναλάβουν το παιδί αυτό είναι ότι μιλάμε ρωσικά. Μα είναι έγκλημα να μιλάει κανείς ρωσικά. Αυτό προβάλλουν οι τοπικές αρχές. Πρόεδρος, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά θέματα στην συνέντευξη. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Αυτά που συμβαίνουν στην περίπτωσή μου δεν είναι θέμα ότι έτσι προστατεύεται το παιδί. Δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντά του. Είναι όμως κυρίως θέμα διακρίσεων. Σας παρακαλώ λοιπόν να με βοηθήσετε όσο θα μπορούσατε. Γιατί έχω να κάνω με συμμορία και σας δίνω και αυτή την απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα. Η πρώτη δεν έχει ημερομηνία και η άλλη είναι προχρονολογημένη και με απειλούν ότι όταν επανέλθω στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ θα με συλλάβουν για να δω το παιδί μου. Είναι πολύ σοβαρή απειλή. Μου είπαν ότι αν επιστρέψετε με το παιδί σας θα συλληφθείτε. Και το παιδί σας θα πάει σε θετούς γονείς και θα εξαφανιστεί. Σας παρακαλώ να ε, εξετάσετε το θέμα αυτό από πιο προσεκτικά. Ευχαριστούμε για τη δήλωσή σας, πολύ σημαντική και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, όλο το χρόνο του κόσμου για να το συζητήσουμε μαζί σας. Το καταλαβαίνουμε ότι υποφέρετε κι εσείς και το παιδί σας. Υπάρχουν παρόμοιες υποθέσεις, όχι ακριβώς ίδιες βέβαια με τη δικιά σας και θα ακούσετε και τους άλλους αναφέροντες μέχρι να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σε σχέση με το σημείο αυτό. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής δεν ακούγεται. Ακούστε, δεν μιλάτε με μικρόφωνο και δεν σας ακούμε. Ποιος, όποιος πειράξει το παιδί μου, και μια τρίχα, θα έχει να κάνει με ένα και συγγνώμη που σας τα λέω έτσι. Πρόεδρος, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αφού έχετε υποφέρει τόσο πολύ, θυμώνετε. Έχετε οργή. Είναι κατανοητό. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή, που είναι η κυρία Γκλαζεύσκα. Έχετε το λόγο κύριε Γκλεζεύσκα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στρέφομαι σε εσά για να ζητήσω τη βοήθειά σας εκ μέρους παιδιών που δεν έχουν ε, καμία βοήθεια. Είμαι Πολωνέζα, υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ένας γονιός συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή απευθύνθηκε σε ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να συζητιέται. Δεν πρέπει να μας διώκουν γι' αυτό. Θέλω να βοηθήσω τις δεκάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία ε, ουσιαστικά έχει όμοιρους στο Βρετανικό σύστημα. Αγωνίζομαι κι εγώ δύο χρόνια για την επιστροφή παιδιών. Το σύστημα δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, Απλώς και μόνο θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των υιοθεσιών. Ένας ε, κοινωνικός λειτουργός προσπάθησε δύο φορές να με κάνει να υπογράψω και να συμφωνήσω με χαρτιά υιοθεσία. Με κατηγορούν ότι έχω καταχρηστεί σεξουαλικά το ίδιο μου το παιδί. Έγινα συνεντεύξεις με την αστυνομία. Το παιδί μου ποτέ δεν είπε τίποτα που να μπορούσε να οδηγήσει κάποιον να πιστέψει ότι υπάρχει κάποια αλήθεια στις κατηγορίες αυτές. Παρόλα αυτά, διώκομαι με την κατηγορία αυτή ότι ασέλγησα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες λένε ότι έκαναν προειδοποίησεις, ότι με, μου έστειλαν κοινοποίησεις. Εγώ ποτέ δεν έλαβα τίποτα τέτοιο. Ενημερώθηκα μέρες μετά. Ο πατέρας ε, των παιδιών επίσης εκβιάζεται για να συμφωνήσει να δώσει τα παιδιά. Τα παιδιά επίσης δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε στη μητέρα τους, ε, στον πατέρα τους, ούτε στην οικογένειά τους, τους αρνούνται ακόμα και την υπηκότητά τους. Εγώ ζήτησα τα παιδιά να μπορούν να πάνε στην ε, Πολωνική Εκκλησία και να πηγαίνουν και στο σχολείο μετρικής γλώσσας του Σαββάτου. Το αρνήθηκαν. Με φυλακισμένοι έχουν περισσότερα δικαιώματα. Δεν τους αρνούνται ούτε την ταυτότητά τους, ούτε τις σχέσεις με την οικογένειά τους, ούτε την πολιτιστική τους κληρονομιά, ούτε τη θρησκεία τους. από τότε που είναι στη θετή τους οικογένεια, τα παιδιά είναι πεινασμένα, φοράνε βρώμικα ρούχα. Τίποτα δεν έγινε όταν επέστησα την προσοχή των αρχών σε αυτό. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και η θετή οικογένεια είναι υπεύθυνε για τρομερά ψυχολογικά τραύματα γιατί ανάγκασαν τα παιδιά να κάνουν ψεύτικες δηλώσεις και σε σχέση με τις ασέλγες αυτές τις οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα. Το παιδί μου έφυγε από το σχολείο, το σκασε, γιατί ήθελε να είναι μαζί μου οι αρχές όμως λένε, υποστηρίζουν ότι δεν θέλει να με δει το παιδί. Την τελευταία φορά που τον συνάντησα είπε ότι ήθελε να έρθει να ζήσει μαζί μου. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Και αυτό γιατί προφανώς τον έχουν τιμωρήσει γιατί είπε κάτι που δεν έπρεπε να έχει πει. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με την κόρη μου. Η κοινωνική λειτουργία αρνούνται την επαφή των γονιών με τα παιδιά. Δεν έχω δει τα παιδιά μου τους τελευταίους 7 μήνες. Το δικαστήριο επέτρεψε στον πατέρα να δει τα παιδιά του, αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν το επιτρέπουν αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή από το δικαστήριο, αλλά όχι από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές υπηρεσίες κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τις δικές μου προσπάθειες να έχω τα παιδιά πίσω στην Πολωνία. Με έχουν ε, προσβάλει, ταπεινώσει. Και τέσσερις μήνες αφότου μου τα πήραν, μου είπαν ότι τα ρούχα τους ήταν γεμάτα περιτώματα. ότι υπήρχε δηλητήριο στην τροφή των παιδιών. Το δικαστήριο όμως ήταν πολύ επιλεκτικό όταν έπρεπε να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Και τελικά ευνόησε τις δηλώσεις που έκαναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και όχι τις δικές μου. Ό,τι έγραφα έδωσα εγώ από ανεξάρτητες πηγές απορρίφθηκαν. Έγραφα, το οποία ήταν και ιατρικής φύσεως. Δεν μπορώ να τα δω εγώ. Νομίζω ότι ό,τι έγινε, έγινε κυρίως εξαιτίας της προέλευσής μας. Οι Πολωνοί υποφέρουν από πολιτικές διώξεις και διώξεις στα μέσα ενημέρωσης εξαιτίας των στερεότυπων που ισχύουν, εξαιτίας των παραδόσεων. Οι πολωνικές οικογένειες έχουν απειλές που τους γίνονται και υποφέρουν από διακρίσεις και ρατσιστικές επιθέσεις. Χωρίς κανένα λόγο οι πολωνικές οικογένειες διαπιστώνουν ότι χάνουν τα παιδιά τους, τους τα παίρνουν. Στην αρχή συγκέντρωνα αποδεικτικά στοιχεία, έπαιρνα φωτογραφίες, ρωτούσα, προσπαθούσα να βρω στήριξη. Τώρα όμως ξέρω ότι δεν πρόκειται για τη δικαιοσύνη. Τώρα ξέρω ότι πρόκειται απλώς και μόνο για την αμάυρωση των ονόματος των ανθρώπων και για την στέρηση του δικαιώματος στους γονείς να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Με κατηγορούν για ένα σωρό πράγματα. Βάζοντας λόγια στα στόματα των παιδιών μου. Η κοινωνική λειτουργή δεν θα έπρεπε να αντιδρούν έτσι και να μισεύονται τα συμφέροντα των παιδιών και των γονιών. Δυστυχώς όμως το σύστημα δεν υπόκειται σε επαρκή έλεγχο και γίνονται καταχρήσεις. Δεν είναι τελικά τα δικαστήρια αυτά τα οποία αποφασίζουν, αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και κάνω έκκληση σε εσά να εξετάσετε αυτήν την προσωπική τραγωδία και να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους. Ευχαριστώ. Thank for having Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κυρίως που είχατε το κουράγιο να, μας, να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας, που πραγματικά ραγίζει καρδιές. Επόμενη Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι αρχές της ε, Λιθουανίας, ε, λέει η αδελφή μου την οποία εκπροσωπώ, μου πήραν το διαβατήριο και έτσι μπόρεσα να έρθω να παρουσιάσω την ε, αναφορά μου στην Επιτροπή Αναφερών. Ο γιος μου που είναι Λιτωνός ε, υπήκος, γεννήθηκε το 2007, το 2011, ε, χωρίς απόφαση δικαστηρίου, τον απήγαγαν ε, το Σεπτέμβριο, μάλλον το 2013 πήχθη από την τουαλέτα και δεν υπήρχε ούτε διερμηνέας, ούτε φορείο. Το παιδί φώναζε στα αγγλικά «Θέλω να ζήσω με τη μαμά μου». Η Σάλεν Βαρμίνεν, η κοινωνική λειτουργός, δεν είναι καταχωρισμένη στο επαγγελματικό μητρό κοινωνικών λειτουργών. Απειλήθηκε η μητέρα και το παιδί της ε, ότι θα, τους, ε, θα την εγκλήσουν κυρίως ε, εκείνη στη φυλακή. Το Σεπτέμβριο του 2013, όπως σας είπα, απήχθη το παιδί και έκτοτε είναι μακριά από το σπίτι του. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στο δημοτικό το 2013 λόγω του ότι λείπουν θέσεις στα σχολεία στο Μπραντ. Υπήρχε προγραμματισμός αυτής της επίθεσης ε, κατά του παιδιού εμείς ε, το μάθαμε αυτό, η μητέρα και η γιαγιά δέχτηκαν την επίθεση, απήχθησαν για 24 ώρες. Η μητέρα και η γιαγιά αντιμετώπισαν πλασματικές κατηγορίες ότι δίθεν επιτέθηκαν σε έξι αστυνομικούς. Ε, δεν υπέγραψα καμία ε, αναφορά, λέει η μητέρα, ε, με βάση την τρέχουσα νομοθετική, λιθουανική νομοθεσία, τα παιδιά ζουν πάντα με τις μητέρες τους. Στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά από τρεις ημέρες από την απογωγή του παιδιού μου, το παιδί μου μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αναφέρθηκαν λάθος στοιχεία για τη μητέρα του και στη μητέρα του αναφέρθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία εκδίκαση της υπόθεσης οι κοινωνικές υπηρεσίες ισχυρίστηκαν ότι το πατέρα του κακοποιεί, ο πατέρας του κακοποιεί το παιδί. Η μητέρα και το παιδί ψυχιατρικά είναι υγιείς, αλλά από τότε που υπήρξε η πρώτη απόφαση, οι τοπικές αρχές ε, ταπείνωσαν την μητέρα και την έχουν απειλήσει με εγκλισμό σε ψυχιατρία και σε σοφρονιστικά καταστήματα. Το παιδί ε, πεστράφει στον πατέρα του που το κακοποιεί σεξουαλικά το παιδί μου δεν την χάνει της ε, βέλτιστης δυνατής μεταχείρισης όταν είναι κοντά στο βιολογικό του πατέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες της ε, Λιθουανίας ε, παρουσίασαν παραποιημένα έγγραφα στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και τα έγγραφα αυτά ε, κρίθηκαν παράτυπα από Λιθουανούς νομικούς Το παιδί όμως, ε, όπως σας είπα, μετά από ένα χρόνο σε ανάδοχη οικογένεια επιστράφηκε στον πατέρα του ε, παρότι η μητέρα είχε ζητήσει την προστασία από τον πατέρα από τις λιθουανικές αρχές. Οι λιθουανικές ε, αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει αυτή η κακοποίηση από τον πατέρα έγιναν εξετάσεις ε, ιατροδικαστικές, ε, το παιδί κατέθεσε στην αστυνομία, στη Λιθουανία αλλά και στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και υπάρχουν αποδείξεις ε, για την κακοποίηση από τον πατέρα. Εξάλλου ο πατέρας έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό. Οι Λιθουανοί ψυχολόγοι κατέληξαν ότι ο πατέρας είναι ψυχοπαθής. Το παιδί μου ζητάει να σωθεί από τον πατέρα του, από την κακοποίηση, αλλά κανείς δεν τον ακούει. Το παιδί μου λέει ότι είναι ευτυχισμένο με τη μητέρα του, αλλά κανείς δεν μοιάζει να κατανοεί τον πόνο του. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αγνόησαν την επιθυμία του παιδιού, το μετέφεραν στη Λουρατανία, το παρέδωσαν στον ψυχοπαθή πατέρα του έδωσαν δυνατότητα να το κακοποιήσει περαιτέρω και η υγεία του παιδιού όταν ε, απομακρύνθηκε από τη μητέρα του επιδεινώθηκε σοβαρά. Το δικαστήριο δυστυχώς απαγόρεψε στη μητέρα να μιλάει για την τραγωδία της. Οι αρχές της Μεγάλης Βρετανίας παραβίασαν την απαγόρευση διακριτικής μεταχείριση λόγω γλώσσας και ε, των έμεσων διακρίσεων λόγω εθνοτικής προέλευσης και ηθαγένειας. Διακόπτη Πρόεδρος, ε, συγγνώμη κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι αυτά που διαβάζετε είναι μακροσκελή θα έλεγα, αλλά μήπως μπορείτε να φτάσετε κάπως στο τέλος αυτής της επιστολής. Θέλω να πω ότι παραδιάστηκαν πολλά άρθρα ε, πολλά δικαιώματα του παιδιού Το παιδί το άρπαξαν από μια οικογένεια που το αγαπούσε και το έδωσαν σε ανάδοχη οικογένεια αλκοολικών. και από τους αλκοολικούς επεστράφει στον ε, βιολογικό του πατέρα που το κακοποιεί. Πρόεδρος, λυπάμαι πάρα πολύ που σας διακόπτω όλους, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είστε συναισθηματικά φορτισμένοι, αλλά πιστέψτε με, πρέπει να προχωρήσουμε. Και τώρα θα δώσετε το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούσαμε. Yes, thank you very much. I have... Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους αναφέροντες και σας ευχαριστώ που κάνατε όλη αυτή την προσπάθεια να έρθετε στις Βρυξέλλες για να μας ενημερώσετε για τις ε, οδυνηρές εμπειρίες σας και λυπάμαι για τις ε, ε, απίθμενες δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε και καταλαβαίνω πόσο όλα αυτά σας τυραννούν. Όπως είπα και στην κυρία Μακνίου, δεν θα σας πω τις συνηθισμένες γενικολογίες για έλλειψη αρμοδιότητας. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιους αναφέρονται σαν, όχι όλους βέβαια, είναι ότι οι αποφάσεις των κοινωνικών υπηρεσιών μπορούν να αμφισβητηθούν. Τα δικαστήρια στον Αμένο Βασίλειο μπορούν ενδεχομένως να ακυρώσουν αποφάσεις ε, κυβερνητικών τοπικών αρχών αν είναι πεπισμένα ότι αυτή η απόφαση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παιδιού και τους γονείς του. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε αυτές τις ε, νομικές και υπάρχει γραφείο συμβουλών για του πολίτε του Ηνωμένου Βασίλειου που μπορεί επίση να σα βοηθήσει. Θα σα δώσω τα αναγκαία στοιχεία όπω είπαν οι Βρετανικές αρχέ στην επιστολή την οποία ανέφερε και η οποία διανεμήθη σήμερα με βάση το νόμο για τα παιδιά που ε, είναι το πλαίσιο για το σύστημα προστασία. οι τοπικέ αρχέ πρώτα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει ένα παιδί να επιστρέψει στους γονείς του. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει το παιδί αυτό να ε, δοθεί σε ένα μέλος της ευρύτερης οικογένειας ε, του παιδιού γιατί είναι καλύτερα να ζει με το παιδί με κάποιον που ε, γνωρίζει ήδη και μόνο αν αυτό δεν επιτύχει θα πρέπει να δοθεί σε άλλους. Θα είμαστε σε επαφή με τις Βρετανικές Αρχές για τα θέματα αυτά και καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχει δυνατότητα η Επιτροπή σας να κάνει μια επίσκεψη ε, ενημέρωσης για να έχει καλύτερη εικόνα, πληρέστερη, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που θέλω να προσθέσω, το είπα και προηγουμένως, είναι μετά από τη συνάντηση της Επιτροπής Αναφορών τον Μάρτιο, ε, κάναμε ήδη ε, μια, θέλουμε ήδη να κάνουμε μια μελέτη για την κατάσταση προστασία των παιδιών στα κράτη-μέλη και να δούμε πώ είναι δυνατόν να προστατεύσουμε καλύτερα τα συμφέροντά του σε περιπτώσει που καλύπτουν και υιοθεσία και επιμέλεια. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα δημοσιευθούν και με βάση αυτή την εργασία θα διατυπώσουμε νωρίς στις αρχές του 2015 κατευθύνες γραμμές που να βασίζονται σε μια προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών για να βοηθήσουμε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών. Πρέπει να υπερβούμε τις υπάρχουσες διαδικασίες και δομές, να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και ότι προστατεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις γνώσεις μας για τον τομέα αυτό. Πρόσφατα η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες για περισσότερο προσωπικό στον τομέα αυτό η πρώτη μας προτεραιότητα και δεν μπορώ να την υπογραμμίσω αρκετά είναι να βασιζόμαστε στη λήψη υπόψη των συμφερόντων των παιδιών και στα δικαιώματά τους. Και επίσης αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα του παιδιού να γίνει ακουστή η άποψή του. Αυτό πρέπει να είναι βασικό σε θέματα επιμέλειας όπως αυτά που συζητάτε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Μόνο ο κύριος Σάκη είναι στο κατάλογο μιλητών. Να του δώσω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος. Θα προσπαθήσω. Πρώτον. Βλέπω ότι δεν έχουμε μεμονωμένα προβλήματα, αλλά υπάρχουν πολλά. Άρα υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Η σύστασή μου λοιπόν προς όλους μας και την Επιτροπή είναι να ενημερώσουμε τον κύριο Τίμερμανς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι εδώ διαπιστώνουμε σοβαρό πρόβλημα. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την ε, διαμεσολαβήτρια εάν έχουν ε, πληροφόρηση ή παρόμοιες περιπτώσεις και να την καλέσουμε για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε και να ζητήσουμε την Επιτροπή να μας υποβάλλει μια ανάλυση της κατάστασης. Αυτά είναι ε, βήματα συνεκτικά. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα νέο νομοθέτημα, ένα νέο σύστημα για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Διότι διαπιστώνω ότι να συνεχιστεί ως έχει η συζήτηση, να δηλαδή ακούσουμε και για άλλες περιπτώσεις στο μέλλον, δεν επαρκεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πιο συστηματικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και πώς τώρα μπορώ να κλείσω τη συζήτηση. Ως εξή. Πρώτα απ' όλα οι αναφορές παραμένουν ανοιχτές. Αυτό είναι αναγκαίο. Πρέπει σε βάθος να εξετάσουμε τα θέματα και παρακαλούμε την γραμματεία μας να συνεργαστεί με τις νομοθετικές επιτροπές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι οι επιτροπές ε, Τζούρι και Λίμπε έχουν ζητήσει μια μελέτη για θέματα απαγωγών παιδιών διαμεθοριακά. Αυτή η έκθεση θα υποβληθεί σύντομα στην ε, Τζούρι και τη Λίμπε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καλέσουμε τη γραμματεία μας να απευθυνθεί σε αυτές τις δύο επιτροπές και να μας καλέσουν και εμάς στην παρουσίαση. Γιατί ακούσαμε σήμερα για διάφορες περιπτώσεις και ακούσαμε και τι μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σύντομα και τις κατευθύνες γραμμές και τα αποτελέσματα της έρευνας της ε, υπηρεσίας θεμελιδών δικαιωμάτων. Ήδη σήμερα είπαμε ότι θα καλέσουμε τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαντ στην ε, Επιτροπή μας. Θαυμάσιο θέμα λοιπόν αυτό να είναι στην σε διάταξη όταν θα έρθει στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτήν την επιστολή. Είναι απαράδεκτο. Ένας Ευρωπαίος πολίτης να απειλείται αν επιχειρεί απλώ να ασκήσει το δικαίωμά του να υποβάλει αναφορά. Είναι απαράδεκτο, δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ, απολύτω ποτέ. Άρα πρέπει να γράψουμε στι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου και να υιοθετήσουμε και τα άλλα μέτρα. Η κυρία Ντανόκα. Ναι, ναι, μα και εγώ ήθελα να γράψουμε αυτή την επιστολή. Αλλά είχαμε και την πρόταση από κάποιους που είπανε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αποστολή ενημέρωσης και εξέβρεση στοιχείων. Μα αυτό θα το συζητήσουν οι πρόεδρος, λέει, οι συντονιστές. Έχουμε πολλά θέματα, πρέπει να είμαστε πολύ περιοριστικοί. Πολλά θέματα που εκκρεμούν. Νομίζω ότι αν δράσουμε με σωστό τρόπο και συνεργαστούμε με τις νομοθετικές επιτροπές στενά, θα επιτύχουμε περισσότερα. Για να αντιμετωπίσουμε την ουσία των θεμάτων. Εάν λοιπόν έρθει εδώ ενώπιόν μα, σύντομα ο κύριο Τίμερμαν, Έχουμε πολλά θέματα που μπορούμε να του θέσουμε και αυτό οπωσδήποτε θα ήταν από τα κυριότερα. Είναι αντιπρόεδρο τη της Επιτροπή. Επιτροπής. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και πρέπει να λήξει όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Όπω είπε ένας συνάδελφος, έχουμε ακούσει και σε άλλε περιπτώσει και για άλλε περιπτώσει σε τρίτες χώρε, αλλά στην Ένωση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Οπωσδήποτε θα έπρεπε. Συμφωνείτε επί των προτάσεων αυτών, παρακαλώ. Η κυρία Σμίτσι Κάθε διαμαρτυρία που ακούσαμε σήμερα είναι σημαντική, αλλά εφόσον μιλάμε για παιδιά, δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνουν όλα αυτά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει εδώ ο κύριος ε, Τίμερμαντς. Γι' αυτό προτείνω Ναι, μεν όλα τα θέματα που μας αφορούν είναι σημαντικά και είναι πολύ δύσκολο αυτό που επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Τα προβλήματα για τα οποία ακούσαμε σήμερα που έχουν να κάνουν με παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν. Κάθε μέρα που περνάει είναι άλλη μια μέρα τραγωδίας για τα παιδιά, για τους γονείς επίσης, για άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Γι' αυτό θα πρότεινα Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ιδρύσουμε μια υποεπιτροπή που να ασχολείται μόνο με θέματα παιδιών. Θέματα που είναι όντως πρωταρχικά και δεν μπορούν να περιμένουν. Δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί τέτοια πρόταση, αν έχει ήδη προταθεί παλιότερα, αλλά πιστεύω ότι τα προβλήματα αυτά θα μας απασχολούσαν κάθε μέρα αν είχαμε μια αρμόδια επιτροπή. Τα παιδιά δεν μπορούν να συγκριθούν με το θόρυβο και την ηχορύπανση και το περιβάλλον. Τα παιδιά όμως δεν μπορούν να περιμένουν. Όπως σωστά είπατε, λέει η πρόεδρος, κάθε μέρα που συνεχίζουν τα παιδιά αυτά να είναι μακριά από τους γονείς τους, ε, είναι μια χαμένη μέρα και για ένα παιδί μια μέρα είναι σαν μήνας για ενήλικα. Μα ήδη πήρα μια απόφαση. Είπαμε ότι θα μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα με ταχύτατη διαδικασία. Όλοι συμφωνήσαμε. Όλοι λοιπόν συμφωνούν ότι έχουμε προχωρήσει. Έχουμε προχωρήσει. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, δικηγόρος ε, πρέπει να σχώ σχολήθηκα με το οικογενικό δίκαιο. Κοιτάξτε, η ιδιορυθμία δεν είναι ότι ε, τσακώνονται οι άνθρωποι, αλλά ότι εδώ πρόκειται για το παιδί. Και στην περίπτωση του παιδιού δεν μπορεί κανείς να προβαίνει σε ε, συμβασμούς, συν το ότι υπάρχει συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Όμως, να προσέξουμε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ε, το θέμα των παιδιών εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Και εδώ υπάρχουν τρεις δυνατότητες είτε, ε, και ε, μετά και άλλη μια περίπτωση, είτε έχουμε ευρωπαϊκή νομολογία, είτε η δυνατότητα κάποιος να υφίσταται διάκριση από το εθνικό σύστημα, μόνο και μόνο διότι έχει διαφορετική ηθαγένεια από το κράτος ε, όπου διαδραματίζεται η υπόθεση. Ε, δηλαδή αν θέλετε εδώ η δυνατότητα είναι το ενωσιακό δίκαιο. Και το τρίτο που υπάρχει είναι ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για όλα αυτά όμως υπάρχουν δικαστήρια και κατά δική μου άποψη θα ήταν σκοπιμότερο να απευθυνθεί κανείς στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβουργό και εκεί να υπάρχει ε, επιταχυμένη διαδικασία για θέματα παιδιών. Διότι εκεί ακριβώς λαμβάνονται αποφάσεις για την ευημερία των παιδιών. Το λέω αυτό εμείς είμαστε αρμόδιοι για θέματα επιμέλειας ε, παιδιών, όμως σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο για τέτοιου είδους θέματα. Σωστά είπατε κυρία Πρόεδρε ότι ραγίζει η καρδιά μας και στανόμαστε όλη την κατάσταση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να επιταχύνουμε ιδιαίτερα, να μιλήσουμε με τον κύριο Τίντεμαρς ο οποίος πρέπει να γνωρίζει και τα όρια που υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όσο και αν είναι τραγικό. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα σε κανένα κράτος μέλος όπου οι γονείς που βρίσκονται σε διάσταση να είναι ικανοποιημένοι με την απόφαση που λαμβάνει το δικαστήριο. Δυστυχώς αυτό δεν υφίσταται. Πρόεδρος, Πολύ ωραία. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να επαναλάβω, να ανακεφαλαίωσω αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Δηλαδή εμεί από πλευρά γραμματεία θα απευθυντούμε σε άλλε αρμόδιε επιτροπέ ε, για να δούμε τι ακριβώς υφίσταται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικών προτάσεων. Και μετά θα καλέσουμε τον κύριο Τίμερμανς, θα συζητήσουμε μαζί του, θα απευθυνθούμε και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών που έχουν ήδη εκπονήσει μια μελέτη για την απαγωγή παιδιών μεταξύ άλλων. Αυτά θα τα παρουσιάσουν στο πλαίσιο μιας ακρόασης και αυτό τον δρόμο θα ακολουθήσουμε παράλληλα με μια επιστολή που θα στείλουμε στις Βρετανικές Αρχές επισημένοντας το δικαίωμα αναφοράς και το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν απειλέ στην περίπτωση που κάποιο ασκεί το δικαίωμά του αυτού. Η σιωπή σα ε, φαντάζομαι σημαίνει συνένεση. Κατόπιν τούτου ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που αφορά τον ε, κύριο Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο. Σωρίσατε. Ε. Ευχαριστώ. Όλα είναι για σας. Τι παντάμε. Okay, good evening. Ε, this petition... Καλησπέρα. Πρόκειται για την παραφίαση του δικαιώματος επιμέλειας που έχει να κάνει με δύο χώρες μέλη. Οι γη μου ζούσαν στην Κύπρο το 2010 και τους απήγαγε η μητέρα τους. με τη στήριξη των εθνικών αρχών, όπως θα σας εξηγήσω αργότερα, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και βρίσκονται σε τρίτη χώρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό χωρίς τη βοήθεια των εθνικών αρχών της Κύπρου. Από τις επαφές, ε, ή μάλλον οι επαφές ειδικές με τα παιδιά έκτοτε έχουν διακοπεί. Τα παιδιά έχουν την ελληνική υπηκότητα και σύμφωνα με τον Ηνωμένο Βασίλειο κατοικούν στην Ελλάδα. Η μητέρα τους είναι Ουγγαρέζα, αλλά έχει και Βρετανικό διαβατήριο. Και έτσι μπορούσαν και τα παιδιά να έχουν Βρετανικό διαβατήριο εξαιτία τη σύνδεση αυτή τη μητέρα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα είχε γίνει αυτό χωρίς την συμμετοχή των Βρετανικών Εθνικών Αρχών που έδωσαν τα διαβατήρια στη μητέρα. Ενώ γνώριζαν τις δυσκολίες που υπήρχαν, γνώριζαν ότι υπήρχε δικαστικό θέμα για την επιμέλεια των παιδιών στην Ελλάδα, που έχει και το δικαίωμα να αποφασίσει για αυτά. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι πίσω από κλειστές πόρτες, στο Λονδίνο, στην Υπουργείο Εξωτερικών, Πρωθυπουργού, αποφάσισαν το θέμα να το πάρουν από τα ελληνικά δικαστήρια και να το δικάσουν οι ίδιοι. Χωρίς βέβαια δικαστές, χωρίς δικηγόρους, χωρίς να χάσουν χρόνο, χωρίς μάρτυρες και αποφάσισαν ποιος τελικά από, τα δύο, από τους δύο γονείς θα έχει την επιμέλεια. Πού θα ζήσουν τα παιδιά και πώς θα μεγαλώσουν. Γνώριζαν ότι ίσως δεν θα μπορούσα να τους ξαναδώ. Η γυναίκα μου μάλιστα πήρε κάποια νομική δράση, ανέλαβε κάποια νομική δράση και έτσι δεν μπορώ μετά από αυτήν να επισκεφτώ τα παιδιά, ούτε εκείνα μπορούν να έρθουν σε μένα. Σύμφωνα με την νομική αυτή απόφαση. Και δεν έχουν καμία επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώρισαν αργότερα το σφάλμα τους και η απάντηση ήταν ότι όταν τους δώσαμε το διαβατήριο στην γυναίκα μου δηλαδή, της είπανε ότι πρέπει να ελέγξει όμως τον νόμο πριν πάρει τα παιδιά και φύγει από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δηλαδή τι είναι αυτό, αυτό θυμίζει ανέκδοτο. Γιατί τώρα τι λένε, λένε μα εμείς τις είπαμε να μην το κάνει. Όσον αφορά τώρα τις Κυπριακές Αρχές, και πάλι εδώ, κάτω από περίεργες συνθήκες, σταμάτησε το διεθνές ένταλμα το οποίο είχε ξεκινήσει κατά της μητέρας μια που το έγκλημα αν θέλετε να το πούμε έτσι έλαβε χώρα στην Κύπρο και μπορούν έτσι να βάλουν τη Eurojust να δραστηριοποιηθεί και να εκδώσουν και διεθνές ένταλμα. Όμως σε 24 ώρες διακόπει η διαδικασία αυτή. Και δεν κατάφερα να αντιστρέψω τη διαδικασία. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, είναι ο πιο σύντομος δρόμος και συμβαίνει δυστυχώς κάθε μήνα στην Κύπρο γιατί υπάρχουν πολλά μεικτά ζευγάρια που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους πίσω. Τώρα εδώ πρέπει να σας πω και δύο λόγια για την περίπτωση αυτή αυτή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν συνυπογράψει τη συνθήκη της Χάγης, οπότε δεν προβλέπονται διαδικασίες για να επιστρέψουν τα παιδιά. Εδώ πέρα εξετάζουμε την ε, υπόθεση βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Παρόλο που το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το απέκρυψε. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως το αναγνώρισε όταν εξέτασε την ε, δικιά μου την καταγγελία σε βάρος της Κύπρου και όταν απάντησα στις 19 Σεπτεμβρίου, απάντηση που έστειλα και στην γραμματεία, έχω συμπεριλάβει και επιστολές και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου το παραδέχονται. Τα οικογενικά δικαστήρια στην Ελλάδα ε, όντω κατέληξαν στο ότι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα. Ε, ο ΔΕ Υπουργό Δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε ότι η υπόθεση αυτή εξετάζεται βάσει κανονισμών και είναι θέμα Βρετανικής νομοθεσίας και Βρετανικών νόμων σε δικαστική όμως συνεργασία για οικογενειακά ζητήματα. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να βρει και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν εκεί κάποια στοιχεία και η δικιά μου βέβαια είναι μια συγκεκριμένη. Αν πάτε στο μενού θα το δείτε και η επιστολή που έστειλα εγώ είναι η ίδια η επιστολή που έστειλα και στην Επιτροπή σας Αναφορών με διαφορά μιας εβδομάδας. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνωρίζει πώς χειριζόμαστε το θέμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νιοθετεί τη θέση ότι η έκδοση διαβατηρίων δεν είναι θέμα κοινοτικού δικαίωμα. Το θέμα δεν είναι το διαβατήριο αυτό καθ' αυτό, είναι ότι ως πατέρας που έχω την κυδαιμονία ακόμα, έχω το δικαίωμα να αποφασίσω πού θα κατοικήσουν τα παιδιά μου βάσει του άρθρου 249 του κανονισμού του 2003. Και οι Βρετανικές αρχές δίνοντας ταξιδιωτικά έγγραφα στην μητέρα, της δίνει το δικαίωμα να απομακρύνει τα παιδιά από μια χώρα μέλος και μακριά από χώρα όπου μπορεί να υπάρξει δικαστική διαδικασία. Πριν μιλούσαμε για το συμφέρον των παιδιών. Πολύ πρόσφατα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ετοίμασε μια μεγάλη μελέτη με απόφαση του 2010. Στην παράγραφο 16 το δικαστήριο αποφάσισε σε συνδυασμό με το σημείο 13 του κανονισμού ότι αναγνωρίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και οι διατάξεις του κανονισμού αυτού δεν μπορούν να τύχουν ερμηνείας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη το θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού το οποίο σημαίνει το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Οι Βρετανικές αρχές λοιπόν αλλά και οι Κυπριακές αρχές αποφάσισαν από μόνε του ότι το καλύτερο συμφέρον του παιδιού είναι να μην συναντάει τον πατέρα του. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για πόσο ακριβείς ήσταν και ευχαριστώ επίση και για την παρουσίαση με διαφάνειε. Έτσι είναι ευκολότερο να παρακολουθήσουμε την επιχειρηματολογία σα ε, για όλα αυτά βέβαια τα οποία, από τα οποία υποφέρετε. Να δώσω το λόγο απευθεία στην Επιτροπή. Είναι η Κλέρα Νέσ Μαγνία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρούσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρον είναι ιδιαίτερα οδυνηρή. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε με πολύ προσοχή τα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρον. Επίσης τον ακούσαμε, τον συναντήσαμε δύο φορές για την κατάσταση που αντιμετωπίζει. Έχουμε κάθε κατανόηση για το πόσο υποφέρει που δεν μπορεί πια να έρθει σε επαφή να δει τα παιδιά του. Εξετάσαμε όλες τις πλευρές και όλα τα στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα όσα επράχθησαν στην Κύπρο και η κατάληξή μας είναι ότι από όλα τα στοιχεία αυτά δεν βλέπουμε παραλήψεις από πλευράς των κρατών μελών έναντι της νομοθεσίας της Ένωσης. Βεβαίως, σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον αναφέροντα να ανακτήσει την επαφή με τα παιδιά του. Η δυσχέρεια είναι ότι τα παιδιά του είναι τώρα σε τρίτη χώρα εκτός Ένωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα έναντι ενός τρίτου κράτους. Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως προσπαθεί να ενισχύσει την ε, συνεργασία σε θέματα οικογενειακού δικαίου με τα τρίτα κράτη με βάση πολυμερή πολυμερείς δυνατότητες που έχουμε, για παράδειγμα τη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα θέματα αστικού δικαίου των ε, διεθνών απαγωγών παιδιών και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα αλλά δεν συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε κάθε κατανόηση, ακούσαμε και σήμερα τον αναφέροντα να τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές οι αρχές δηλαδή ενός κράτους μέλους είχαν κληθεί να αποφασίσουν για την επιμέλεια των γονέων επί των παιδιών. Αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ στην Επιτροπή σας και στον αναφέροντα είναι ότι αν αυτή η οδός δεν επιτρέψει να βελτιωθεί ουσιοδός η κατάσταση θα έπρεπε να διερευνήσει ο αναφέρον τη δυνατότητα να ζητήσει αρρωγή μέσω της διπλωματικής οδού για να επιχειρήσει να ξεμπλοκάρει την κατάσταση συγκεκριμένα. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα εκ νέου να έρθει σε επαφή με τα παιδιά του. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο σε όσους συναδέλφους θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Η Ελεονόρα Εύη. Ευχαριστώ πολύ. Οι περιπτώσεις ε, για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα το απόγευμα είναι περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολες, σοβαρές και νομίζω αυτό το οποίο προέκυψε ξεκάθαρα είναι ότι είναι απαραίτητο να καλυφθούν κενά που υπάρχουν. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά ξέρετε και αυτό δεν είναι ικανοποιητική απάντηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορούν να υφίστανται τέτοιου είδου καταστάσεις όπου η ζωή αυτών των ανθρώπων κατασπαράσεται από τις ε, διάφορες διοικήσεις κρατών μελών. Πρόκειται εδώ για ζωές, για τους γονείς, για τα παιδιά τα δικαιώματά τους παραβιάζονται. Για μένα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να εμβαθύνουμε σε αυτές τις υποθέσεις και με ακροάσεις, γιατί όχι, αλλά και με ειδικές επιτροπές ερευνητικές για να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις όλων αυτών των προβλημάτων. Και στη τελική ανάλυση και το γραφείο του διαμεσολαβητή για τους ανήλικους και εκεί υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος. Άρα δεν έχει αυτός ε, το επαρκές προσωπικό για να δραστηριοποιηθεί και σε νομικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το δεύτερο θα ήταν μια πολύ σημαντική στήριξη των ε, αναφερόντων και των ε, θυγόμενων. Είπα ότι συμφωνώ να υπάρξει μία δημόσια κρόση για αυτή τη συμφωνία τη Βρυξέλλες 2, άρα δηλαδή είναι σαφές ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι, αναφορές με για να περιμένουμε το αποτέλεσμα των δημόσιων διαβουλεύσεων. Αυτό το οποίο επίσης είναι σαφές και που πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη είναι, αυτά είναι θέματα δικαστικής αρμοδιότητας και νομίζω ότι θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Ο κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, όπου δεν μπορούμε να τις χειριστούμε εύκολα. Είναι δύσκολες ε, περιπτώσεις, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιο συγκεκριμένα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στην Επιτροπή για το θέμα της αναθεώρησης της Συμφωνίας Βρυξέλλες 2α. Μπορώ κάλλιστα να φανταστώ ότι για να αποφύγουμε κακοποιήσεις, ε, τέτοιου είδου περιπτώσει να περιμένουμε μια δεσμευτική δήλωση εκ μέρου των κρατών μελών, έτσι ώστε περιπτώσει όπου υπάρχουν διαζύγια, χωρισμένοι γονεί που προέρχονται από δύο διαφορετικά κράτη-μέλη, πράγματι είναι ένα απαραίτητο να υπάρχουν δύο υπογραφέ για την έκδοση διαβατηρίου. Και στην περίπτωση όπου υπάρχει μόνο μία υπογραφή και ο άλλο αρνείται, τότε να μπορεί να αντικατασταθεί η δεύτερη υπογραφή μόνο από δικαστή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσει όπου πράγματι πράγματι κολλείεται ο γονέας να δώσει την υπογραφή του, εκεί να μπορεί να παρεμβαίνει ο δικαστής. Δεύτερον, στην περίπτωση της ε, απομάκρυνσης παιδιών με τη Συμφωνία Βρυξέλλες 2 να υπάρξει μια συμφωνία ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις τα εντάλματα, διεθνή εντάλματα σύλληψης να εκδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κυρίως στις περιπτώσεις ε, κρατών με τις οποίες δεν έχουμε συνάψει συμφωνία επαναπατρισμού. Δεν εννοώ απαραίτητα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ξέρετε υπάρχει κάποια σχέση με χώρες που δεν έχουν υπογράψει αυτές οι συμφωνίες επαναπατρισμού, δηλαδή ε, είναι χώρες ε, όπου πηγαίνει κανείς γιατί πιστεύει ότι θα τον αφήσουν ήσυχο. Όμως πρέπει ως το πράττουν αυτό να γνωρίζουν ότι αν θέλουν να επιστρέψουν θα εκτεθούν, ε, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση όπου ε, θα πρέπει να παραπέμψουμε στον τον αναφέροντα ή να το επισημάνουμε τη δουλειά και το γραφείο της κυρίας Μαγκίνες που επιλαμβάνεται ιδιαίτερα της ε, εκπαίδευσης και της ανατροφής των παιδιών. Ξέρετε, έτσι με μικρά βήματα, μικρή διπλωματία, νομίζω ότι κάτι μπορείτε να πετύχετε. Και εξάλλου, κυρία Πρόεδρε, μετά τη συνεδρίαση, αν μου επιτρέπετε, κατηδίαν να δώσω και μία μικρή συμβουλή για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ε, κάποια πρόοδος, αλλά αυτό κατηδίαν. Θα ήταν όντως πολύ χρήσιμο. Μια στιγμή. Θα δώσω το λόγο σε άλλον ένα συνάδελφο και μετά εσείς. Έτσι κάνουμε συνήθως. Σύμφωνοι. Ωραία. Η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνουμε μια πρόταση σε σχέση με την αναφορά του κύριου Ιαννόπολου. Είναι να μένει ανοιχτή η αναφορά και να δούμε και αυτά τα ζητήματα στην ακρόση που τα κάνουμε. Ευχαριστώ. Excellent. And by that... Βεβαίως. Τώρα θα δώσω το λόγο σε εσάς κύριε Γιαννόπουλε. Και πάλι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Έντελμα μπορεί με τη βοήθεια της Eurojust να εκτελεστεί. Η Eurojust με την εντολή που είχε το 2009 μπορούσε να φροντίσει για την εκτέλεση του εντάλματος. Η μονάδα της Eurojust για την προστασία των παιδιών δεν μπορεί να ανοίξει έρευνα παρά μόνο εφόσον τη ζητηθεί από χώρα μέλος. Οι Έλληνες εισαγγελείς στο υψηλότερο επίπεδο δεν μπορούν να ανοίξουν μια υπόθεση γιατί ο χώρος που έλαβε χώρα το έγκλημα δεν ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν συμφωνεί να προχωρήσει στις διαδικασίες σε σχέση με το ένταλμα αυτό και αυτό είναι το σκανδαλώδες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα διαβατήρια χρειάζεται μία υπογραφή. Δεν μπορώ να πάω σε ελληνικό δικαστήριο και να ζητήσω να αποσύρουν διαβατήριο που έχει εκδώσει άλλη χώρα μέλο. Δεν μπορώ να πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί τα παιδιά δεν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε δεν υπάρχει καμία διαδικασία που μπορώ να αναλάβω για να αρθεί το δικαίωμα στα διαβατήρια αυτά. Μόνο η Ευρώπη μπορεί να ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να άρει τα διαβατήρια αυτά. Όσον αφορά τώρα την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, όντως συναντηθήκαμε δύο φορές. Η δεύτερη αναφορά, η αναφορά μου ήταν κατά της Κύπρου, επειδή παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο και τις δικαστικές αποφάσεις όπου απευθύνθηκα για έκτακτα μέτρα. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με άλλες αρχές που δεν αναγνωρίζουν ότι με τον κανονισμό πρέπει να διαθετηθεί αυτή η υπόθεση. Δεν δέχονται ότι η Ελλάδα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία και δεν δέχονται τον ορισμό της απαγωγής που έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Αυτό είναι το περιεχόμενο και η ουσία της αναφοράς αυτής. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλες αναφορές να εξετάσουμε. Τι θα μπορούσε να γίνει. Να στείλουμε επιστολές και, στην Κυπριακή, και στις Κυπριακές Αρχές και στις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά το ένταλμα σύλληψης, όσον αφορά την έγκριση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και όπως και στο προηγούμενο θέμα και εδώ να ζητήσουμε από την γραμματεία να ερευνήσει περισσότερο τι θα μπορούσε να γίνει, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε. Πρέπει λοιπόν πραγματικά όλα αυτά να τα κοιτάξουμε σε βάθος με κάθε τρόπο. Σίγουρα η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κλάου Ζίντζερ. Είσαστε εδώ. Ωραία. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είσαστε πολύ συγκεκριμένος και σύντομος, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι αναβολή 1229 κάθος 2013. Θα, υπο... θα παρουσιαστεί από κοινού με κάποιους άλλους εδώ για πέντε λεπτά. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στη Σύμβαση των Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Εκεί λέει ότι τα κράτη θα σεβαστούν τα δικαιώματα των παιδιών που είναι μακριά από τον ένα και τους δύο γονείς για να έχουν στενή επαφή, απευθείας επαφή και με τους δύο γονείς. Εκτός αν είναι κατά των συμφερών του παιδιού. Το 12 το παιδί του οποίου οι γονείς μένουν σε διαφορετικά κράτη έχει δικαίωμα να έχει τακτική επαφή εκτός αν είναι εξαιρετικές περιπτώσεις στενές προσωπικές επαφές και με τους δύο γονείς. Τώρα να σας πω τα εξή. Έχω τρία έγγραφα που μπορώ να σας δώσω. Το έγγραφο 1 είναι απόφαση δικαστηρίου της Μάλτας που είναι υπό το, το Βρυξέλλες 2α για τα Βρετανικά δικαστήρια και που θα έπρεπε να είναι εκτελεστεί από το Μάρτιο του 2012. Το έγγραφο 2 έκανα αίτηση την 1η Μαΐου 12 για προειδοποίηση με βάση την ε, δικαστική απόφαση και είχε προγραμματιστεί ακρόαση στις 6 Ιουνίου. Έγιναν οι ακροάσεις και αποφασίστηκε να μην υπάρχει επαφή. Σε μία από αυτές τις ακροάσεις μπροστά στο δικαστή κύριο Μόστιν όταν το ρώτησα πώς θα εφαρμόσει το, την ε, Συμφωνία Βρυξέλλες 2α, μου είπε ότι εσείς πρέπει να το οργανώσετε. Αργότερα έστειλα μία αναφορά από ένα νομικό σύμβουλο ότι θα πήγαινα στον Ηνωμένο Βασίλειο για να είμαι σε επαφή με, τις, ε, με, τα, με τα παιδιά. Όμως, οι δικηγόροι της μητέρας ζήτησαν να μου αφαιρθούν τα δικαιώματά μου. Στις 24 Απριλίου 2013 έλαβα μια απόφαση δικαστική του Ενωμένου Βασιλείου που λέει ότι ο πατέρας δεν θα κάνει καμία προσπάθεια να έρθει σε επαφή με το παιδί του. Αυτό έγινε χωρίς να έχω δώσει εγώ καθόλου στοιχεία, χωρίς να έχουν γίνει ισχυριστοί εναντίον μου, ισχυρισμοί εναντίον μου. Ο Βρετανός φορολογούμενος έχει πληρώσει 180.000 λίρες στους δικηγόρους της μητέρας. Και έτσι αντέστρεψαν την απόφαση που υπήρχε για να είμαι εγώ σε επαφή με τα παιδιά μου. Ενώ εγώ ήμουν απόν. Δεν είχα ε, καμία νομική αρρωγή και δεν είχα πλέον πόρους. Ζητώ λοιπόν από την ε, διαμεσολαβήτρια να αναλάβει την ε, αίτησή μου αυτή. Και θέλω να ρωτήσω, Έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμία έρευνα για να δει γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφαρμόζει τι αποφάσει που λαμβάνονται από άλλα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ω επίπτωση, δεν έχω καμία επαφή με το παιδί μου από το 2009 που ήρθε σε επαφή, που, από τότε που πήγε στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. έγιναν τέσσερις μελέτες του διαμεσολαβητή για τι, έγιναν, τι έγινε από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου του Μπρέντ. Αυτό είναι καλό παράδειγμα. Από ό,τι έχω ακούσει, πολλά, ε, πολλοί γονείς δεν μπορούν να απευθυνθούν στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για λόγους φίλου. Δηλαδή, ακόμη και αν ο πατέρας είναι ο κύριος ασκών την επιμέλεια, δεν τον βοηθούν. Και πολύ συχνά μέχρι να υπάρξει δικαστική αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών, έχει χάσει την επαφή ο πατέρας με, τους, ε, με τα παιδιά. Μου είπαν ότι τα, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ενθαρρύνει τα παιδιά να αποφασίζουν εκείνα με ποιον γονιό πρέπει να είναι σε επαφή. Και άλλες αρχές ε, στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν αναπτύξει πρακτικές για να αποφασίζουν παιδιά ακόμη και 8 ετών για το με ποιον γονιό πρέπει να είναι σε επαφή. Ακόμη και 3 ετών παιδιά ερωτώνται επανειλημμένα για το τι πρέπει να γίνει. Και αυτό έχει δημιουργήσει σε καταστροφή πολλών οικογενειών, σε έλλειψη επαφών πολλών παιδιών με τους ε, πατέρες και πολλά άλλα προβλήματα όπως ε, εγκυμοσύνες σε μικρή ηλικία, χρήση ναρκωτικών κτλ. Αγνοούνται τα δικαιώματα των πατέρων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στον ΟΒ Και αυτό δεν βοηθάει την προστασία των συμφερόντων των παιδιών. Καλό την Επιτροπή σας να κάνει μία έρευνα για να δει ποιοι είναι οι λόγοι για τη συστημική αποτυχία του Βρετανικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Ιωάννα Στερτίνσκα. Σωστά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και την δυνατότητα να σχολιάσω. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω γι' αυτό και για την μεταρρύθμιση, την αλλαγή μάλλον στον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Όσον αφορά την αναφορά που εξετάζουμε τώρα, Πιστεύουμε ότι ο αναφέρον γύρει δύο ζητήματα. Το ένα είναι η μία τήρηση της απόφασης 2011 και δεύτερον το άλλο που απορρέει από τα έγγραφα είναι το θέμα της δικαιοδοσίας των ευρωπαϊκών δικαστηρίων να αποφασίσουν για θέματα που έχουν να κάνουν με τη γονική ευθύνη όσον αφορά το παιδί του αναφέροντα. Το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση και είχαμε τη δυνατότητα, χάρη μάλιστα σε επιστολή που εστάλει απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επαναξιολογήσουμε και να ξαναδούμε τα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Και από την τεκμηρίωση αυτή φαίνεται ότι πράγματι η απόφαση αυτή η οποία καταχωρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με απόφαση των ανώτερου δικαστηρίου. Το δικαστήριο ζήτησε από τον αναφέροντα να κάνει αίτηση για την εφαρμογή της απόφασης και από την επόμενη απόφαση διαπιστώνουμε όσον αφορά τις κοινωνικές αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου ότι αναβλήθηκε η επιβολή και ότι ο πατέρας δεν υπέβαλε αίτηση σχετικά με το πώς θέλει να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεύτερον, το θέμα της δικαιοδοσίας που απορρέει επίσης από την τεκμηρίωση που μας υπέβαλε ο αναφέρον. Το επανεξετάσαμε με τις διατάξεις που αναφέρονται τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Ο αναφέρον εξήγησε ότι δεν ήθελε να υποβάλει το παιδί του σε επιπλέον άγχος και το καταλαβαίνουμε αυτό και γι' αυτό και δεν ζήτησε την επιστροφή του. Ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε την δικαιοδοσία της ουσίας το Βρετανικό δικαστήριο και άρχισε τις διαδικασίες όσον αφορά την κυδαιμονία και το δικαίωμα επίσκεψης και επαφής με το παιδί. Μετά από αυτά λοιπόν δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να εντοπίσουμε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Και κατά τη γνώμη μας, στην κατάσταση αυτή για την οποία έχουν την ευθύνη τα Βρετανικά δικαστήρια προκειμένου να αποφασίσουν επί της ουσίας και όσον αφορά την επιβολή της απόφασης της Μάλτας σας είπα ότι τώρα έχει μεταφερθεί και είναι στα χέρια των Βρετανικών δικαστηρίων δεν βοηθούν όλα αυτά τον αναφέροντα για να βελτιώσει τη σχέση του ανάμεσα σε αυτόν και τον γιο του. Μια στενή συνεργασία με το δικαστήριο, με τις τοπικές κοινωνικές αρχές, ίσως θα μπορούσε να δώσει θετικά αποτελέσματα. Και αυτή είναι και συμβουλή που δίνουμε εξάλλου στον αναφέροντα. Έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει σε εθνικό επίπεδο διάφορα μέσα εφόσον τελικά δεν τον ικανοποιήσει η απόφαση. Θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. Όπως ίσως να θυμόσαστε και από την προηγούμενη συνεδρίαση, ήδη το Μάρτιο σας είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει τον κανονισμό Βρυξέλλες 2, που είναι και η κύρια ρύθμιση των οικογενειακών ζητημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε. Ως πρώτο βήμα στην αναθεώρηση αυτή εγκρίναμε μια εφαρμοστική έκθεση η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν το εύρος του κανονισμού και θέματα γάμου και θέματα γονικής ευθύνης και θέματα διαδικασίας επιστροφής παιδιών. Όσον αφορά την επιβολή, κάτι που αφορά και την αναφορά που εξετάζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στην έκθεση αυτή ότι στην πράξη όλοι έχουν να κάνουν με την πραγματική επιβολή των αποφάσεων και υπογραμμίζουμε επίσης ότι η επιβολή αυτή καθεαυτή είναι κάτι που έχει να κάνει με την ομοθεσία του κάθε κράτους. Ο τρόπος επιβολής διαφέρει από χώρα σε χώρα και καταλήξαμε στο ότι αυτό μπορεί να καταλήξει και το είδαμε και από τις διάφορες αναφορές που έχουμε καταλήγει ότι όταν οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η επιβολή της απόφασης. Προκειμένου λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά τις διάφορες υποθέσεις έκανε μια δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του θέρους. Τώρα εξετάζουμε τα αποτελέσματα. Κάπου 200 απαντήσεις είχαμε. Και χαιρόμαστε πολύ για όλα τα σχόλια και τις απαντήσεις που πήραμε και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους γονείς για τα, πραγμάτα, τα προβλήματα στην πράξη που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα με τον κανονισμό αυτών. Έχουμε λοιπόν και την οπτική γωνία των γονιών. Αξιολογούμε τις απαντήσεις λοιπόν αυτή την εποχή. Και σκοπεύουμε να υποβάλουμε πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού μέσα στο 2015. Μπορώ ήδη σήμερα να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά θα καλύπτονται με την αλλαγή που θα γίνει στον κανονισμό αυτόν. Ευχαριστώ. Πολύ καλά νέα αυτά. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε. Τώρα, συζήτηση. Ένας θέλει το λόγο και κλείνω τον κατάλογο ομιλητών, διότι έχουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα να λύσουμε πριν τελειώσουμε. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Βίλαντ. Έχω μία ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την τελευταία φορά ρώτησα κατά πόσον υπάρχουν απευθείας επαφές με, την, το οικείο κράτος μέλος. Κάνατε κάποιες ερωτήσεις στο κράτος μέλος, αυτά τα συμπεριλάβατε στο φακελό σας ή μήπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εκλήθη ποτέ να τοποθετηθεί επί του θέματος. Νομίζω η ε, ερώτηση μπορεί να απαντηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Επιτροπή παρακαλώ. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της ε, προετοιμασίας ε, της αίτηση όπως και της μελέτης αξιολόγησης Πήραμε 28 εκθέσεις από τα κράτη-μέλη και οι πληροφορίες που θα εξάγουμε θα συμπεριληφθούν στη μελέτη οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και θέματα εφαρμογής. Και όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στη μελέτη αντικτύπου. Ο κύριος Βίλαντ, δεν τελείωσα. Αυτή ήταν μια ε, προκατακτική ερώτηση. Άρα δηλαδή η απάντηση είναι όχι. Προφανώς όχι, δεν ήρθατε στην περίπτωση αυτή σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Και θέλω να σας επισημάνω ότι παλαιότερα όταν επρόκειτο για περίπτωση Γερμανίας είχαμε εδώ εκπρόσωπο της γερμανικής ε, κυβέρνησης και τοποθετήθηκε. Εντάξει, σε αυτή τη συνεδρίαση δεν περιμένω απλώς να παρουσιάζεται μια ε, κατάσταση και μετά ε, να ευχαριστούμε θερμά τον αναφέροντα και το όλο θέμα να κλείνει. Αυτό είναι Ελάχιστο, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, επειδή κατέθεσε συγκεκριμένα έγγραφα ο αναφέρον, θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκατε την περίπτωση δεν είναι ικανοποιητικός. Ο αναφέρον ε, δεν προσπάθησε να εκτελέσει ή μάλλον δεν κατέστησαν δυνατές αποφάσεις για να ε, ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα του αναφέροντος. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι αυτό οφείλεται και στα Βρετανικά δικαστήρια στο ότι εξέπνευσε το ένα έτος χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Τρίτον, ο ίδιος ο αναφέρον κατά την ε, προηγούμενη συνεδρίαση είπε και τον και απέδειξε ότι σε χιλιάδες περιπτώσεων μόνο 53 περιπτώσεις ε, αντιμετωπίστηκαν, εξετάστηκαν και λήφθησαν αποφάσεις από αυτόν. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η Συμφωνία Βρυξέλλες 2. Δηλαδή να επιτρέπουμε να εγκρίνεται ένα νομικό κείμενο, αυτό ε, να πρέπει να υπογράφεται από όλα τα κρατημέλη και όμονον αυτό, αλλά μετά να επιτρέπουμε ε, διατάξεις των εθνικών δικαίων να υπονομεύουν το κείμενο το οποίο μόλις έχει υπογραφεί. Μα αν έτσι τα πράγματα, τότε ε, να μην τα ε, ξαναεπαναλάβουμε στο μέλλον. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Η Συμφωνία Βρυξέλλες 2 είναι ισχύον δίκαιο ενωσιακό δίκαιο και ευρωπαϊκό δίκαιο. Και περιμένω από την Επιτροπή να το εφαρμόσει στην πράξη. Επίσης, περιμένω οι ερωτήσεις προς την Κομισιόν να γίνονται όπως πρέπει. Δηλαδή, έχω κάποιες πληροφορίες ότι αυτό δεν λαμβάνει χώρα. Και θέλω να πω στην Πρόεδρο ότι κοιτάξτε, αν κάποιος αναφέρον ε, διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο διοικητική μεταχείρισης της υπόθεσής του, τότε δεν μπορεί η κυρία Ορέλη να απορρίπτει αυτή την διαμαρτυρία, αυτή την προσφυγή λέγοντας ότι εντωμεταξύ εκρεμεί μία αναφορά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και καλό το ότι θα συναντιέστε συχνά με την ε, Ευρωπαία Διαμοσολαβητή και σας παρακαλώ πολύ να το επισημάνετε αυτό που μόλις τώρα σας είπα. Και τελειώνοντας, διαπιστώνοντας ότι η μητέρα του παιδιού πήρε έλαβε βοήθεια, νομική αρρωγή οικονομική για να ε, πληρώσει τους δικηγόρους. Ενώ ο αναφέρον δεν έλαβε καμία απολύτως χρηματοδότηση, διερωτώμε στην περίπτωση αυτή πώς μπορεί να ισχύει η αρχή της δίκαιης δίκης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι για αυτούς τους λόγους πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη δέσμευση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα και αν η υπόθεση αφορά ένα μεγάλο κράτος μέλος και η απόφαση που λαμβάνεται προέρχεται από ένα μικρό κράτος μέλος. Ο κύριος Βίλαντ ε, αναφέρεται σε πολύ σημαντικά θέματα. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Με μία-δύο φράσεις Θέλετε να συνοψίσετε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να σας δώσω το λόγο. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Πρέπει η Κομισιόν να κοιτάξει πολύ προσεκτικά πώς γίνεται αυτή η διεθνή συνεργασία. Και αν δείτε τα αιτήματα που έχω υποβάλει για ενημέρωση, θα δείτε ότι έχω δίκιο. Η εφαρμογή αποφάσεων, η εκτέλεση αποφάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι δυνατή σε κανένα επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη απάντησή σας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μαζί με τα άλλα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει σήμερα πρέπει να τα βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να εργαστούμε γι' αυτό μαζί με τη Γραμματεία και τις αρμόδιες επιτροπές και σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι τώρα που οι Βρυξέλλες 2 είναι υπό αναθεώρηση, μπορούμε να έχουμε πιο προωθημένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για τα θέματα αυτά. Και επίσης θα επιχειρήσω να δω την κυρία Μαγκίνης για το θέμα αυτό. Γιατί είναι η αντιπρόεδρος που είναι αρμόδια για τέτοιου τύπου υποθέσεις, για παιδιά. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να τη συναντήσω για να το συζητήσουμε, όπως πρότεινε ο κύριος Βίλαντ. Αυτές τις δυνατότητες μπορώ να σκεφτώ, αλλά οπωσδήποτε θα μείνει ανοιχτή η αναφορά και θα διαρευνήσουμε κάθε δυνατότητα για να προχωρήσει ο κύριος Βίλαντ. Να καλέσουμε την Κομισιόν με βάση τα νέα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν να απευθυνθεί στο κράτος μέλος και να συζητήσει αυτήν την αναφορά με το κράτος αυτό. Να υπάρξει μια συνέχεια. Πρόεδρος, μα θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Θα καλέσουμε τον κύριο Τίμερο να έρθει εδώ. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τα παιδιά, τους γονείς, τις οικογένειες πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά. Πρέπει να δούμε και πού μπορεί να υπάρχουν ε, κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τα αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Τίμερμανς είναι καλύτερος για καλύτερες ρυθμίσεις, καλύτερη νομοθεσία. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Βίλαντ, κύριε Πρόεδρε. Το σημείο μου είναι, όπως είπα, οι προηγούμενες αναφορές δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτέ γιατί δεν υπήρχε κοινοτική αρμοδιότητα. Μόνο με βάση θέματα γενικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το θέμα αυτό έχουμε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέλω η Κομισιόν να μου πει η υπεύθυνη υπηρεσία, όχι μόνο γενικά ο κ. Τίμερμαντ, θέλω τώρα η Κομισιόν να γράψει στι Βρετανικέ αρχέ και να του θέσει τα ερωτήματα που συζητήσαμε εδώ και να μα ε, παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Α, ναι, πολύ συγκεκριμένο αυτό. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε. Θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή, βεβαίω. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μα είναι τόσο σίγουρο που δεν πρέπει καν να το πούμε. Φυσικά πρέπει να επανέλθει η Κομισιόν. Είπαμε ότι υπήρξε μια διακοπή λόγω της αλλαγής θητείας. Τώρα που έχουμε τη νέα επιτροπή πρέπει κάτι να κάνει. Τελεία. Να περάσω στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το θέμα εντελώς διαφορετικό. Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουμε πέντε διαφορετικές αναφορές. Και έχουμε την τιμή να έχουμε τον Κάρι Γκίβενεν που είναι Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Καλώς ήρθατε. Έχουμε τους αναφερόμενους, τον κύριο Ράιαν, τον κύριο Περμόλες, τη Σάρα Μπαρδία Κονιέ, τον κύριο Μανουέλ Αλτέμιρ Μερχελίνα, Αυτούς. Μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και ίσως η Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει μία απάντηση για όλες, ούτω ώστε στο τέλος της, απα... της μας να έχουμε την απάντησή σας. Για να τελειώσουμε το αργότερο 6.30. Πολ Ράιν, λοιπόν. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, κύριοι ευρωβουλευτές, χαίρομαι που έχω την δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα για να υποστηρίξω την αναφορά, η οποία καλεί για μια ανεξάρτητη εξέταση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων και την απαρχαιωμένη νομική του βάση για να βοηθήσουμε τα παιδιά που θίγονται από τα ελαττώματά του το 2012. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Πολλοί από εσά αναθέτετε την εκπαίδευση των παιδιών σας στα ευρωπαϊκά σχολεία. Και εγώ το έκανα παρόλο που εγώ προσωπικά πλήρωνα διδακτρά. Έχουμε 30.000 παιδιά στα ευρωπαϊκά σχολεία. Και τα ευρωπαϊκά σχολεία θα πρέπει να βοηθούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όπως στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον. Αλλά σήμερα θέλω να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά σχολεία και όχι να βαλτώνουν λόγω της πεπαλαιωμένης νομικής φάσης που σημαίνει δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος. Και γι' αυτό αποτυγχάνουν τα ευρωπαϊκά σχολεία και σέρνονται από τη μία κρίση στην άλλη, βλάπτοντας τους μαθητές. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουν δημιουργηθεί με βάση διακυβερνητική συνθήκη το 1957. Άρα η νομική βάση είναι εκτός των ευρωπαϊκών νομικών νομοθετημάτων. Ναι, τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν υπάγονται στο ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Και κυρίως βεβαίως ε, τα παιδιά αυτά είναι παιδιά εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς είναι δυνατόν, είναι αναχρονιστικό να μην υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εσείς ως Κοινοβούλιο ήδη από το 2011 ζητήσατε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. ομόφωνα ζητήσατε να υπάρξει ριζική αλλαγή της νομικής βάσης. Στο ίδιο ψήφισμα το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η παρούσα νομική βάση έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι σε κατάσταση νομικού κενού. Και κατόπιν υπόθηκε ότι η Κομισιόν είχε κάνει ε, είχε, είχε, είχε ε, υποπέσει σε κακή ε, διοικητική πρακτική. Έτσι είπε ο διαμεσολαβητής. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε τα εθνικά δικαστήρια δεν έχουν καμία δικαιοδοσία. Είναι απαράδεκτος τρόπος αυτολειτουργίας των ευρωπαϊκών σχολείων, νομική έλλειψη βάση στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο ζήτησε να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά παρά την απόφαση και του δικαστηρίου, παρά την απόφαση του διαμεσολαβητή, παρά το ζήτημα ότι πέφτει το επίπεδο των ευρωπαϊκών σχολείων, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Δεν έχει υπάρξει καμία ριζική αλλαγή, συνεχίζεται το νομικό κενό και βλάπτονται τα παιδιά όταν υπάρχουν προβλήματα λοιπόν στα ευρωπαϊκά σχολεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του καθεστώτος. Είναι στην τελική της φάση. Αλλά φαίνεται δεν μπορεί να διορθώσει το νομικό καθεστώς, ούτε καν την πτώση του επίπεδου. Και δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα ουσιαστικό για τα θέματα αυτά στο μέλλον, εάν δεν δράσετε εσείς ως Κοινοβούλιο. Η αναφορά λοιπόν ζητάει να γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη για το τι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν θέλει η Κομισιόν να γίνει κάτι. Παρά το αίτημα του Κοινοβουλίου, παρά την άποψη των γονέων, των παιδιών, του διασαμιλαβητή του δικαστηρίου. Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε, να πάνε στραβά στο ευρωπαϊκό σχολείο. Στη ζωή γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά το βασικό είναι να εξάγονται διδάγματα και να διορθώνεται η κατάσταση. Ε, αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος είναι εντελώς αδιάφοροι έναντι οποιασδήποτε κριτικής και άρα υπάρχει πλήρης αναρχία. Το καλοκαίρι του 2012 αυτά τα σοβαρά σφάλματα συνέβησαν στο θέμα του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, Baccalaureate. Εθίγει και η κόρη μου και πολλοί άλλοι. Ο Επίτροπος Εύκοβιτς ενημέρωσε τον Νοέμβριο του 2013 το Κοινοβούλιο ότι για το Ευρωπαϊκό Μπακαλόρεατ του 2012 η Επιτροπή εκφράζει την ε, λύπη της για τα προβλήματα με τους διαγωνισμούς στα μαθηματικά και τη χημεία. Ζήτησε από τον ε, Γενικό Γραμματέα μια αναλυτική έκθεση που υπέβαλαν οι ορισμένοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και έγιναν κάποιες συστάσεις στις οποίες θα δίδονταν συνέχεια για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να σημειώσετε ότι για τη χημεία τα προβλήματα το 2012 στην πράξη δεν ήταν αντικείμενο καμίας αναλυτικής έκθεσης ε, από το Γενικό Γραμματέα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, δεν έγιναν συστάσεις. Δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Δεν έγινε τίποτα για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ακούστε. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και η Επιτροπή βασίζονται σε μια έκθεση, τη λεγόμενη έκθεση ΡΙΣ 19 12 που θα υποβάλω ως ε, τεκμήριο. Έχει τρεις παραγράφους που κατά τη γνώμη μου είναι άσχετες, ανοησίες είναι στην ουσία, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, είναι ντροπή για τα ευρωπαϊκά σχολεία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελάχιστο μπορώ να πω. Κοιτάξτε αυτές τις τρεις παραγράφους, έκθεση τριών παραγράφων. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας. Γράφηκε από τον εξεταστή, του οποίου η εξετάση ήταν υπό εξέταση. Τι είναι αυτά. Είναι σαν να ψηφίζουν οι γαλοπούλες για το πότε πρέπει να τα Χριστούγεννα. Τι γράφουν λοιπόν αυτοί οι καθηγητές επίσης το 2012 πριν από αυτή την έκθεση προς τις αρχές του σχολείου. Οι καθηγητέ είχαν εκφράσει σοβαρέ ανησυχίε για τα προβλήματα που προέκυψαν. Όμω τα ευρωπαϊκά σχολεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα. Αρνούνται λοιπόν το πρόβλημα. Και έχουν κάνει αυτή, αυτό το πασάλιμα τριών παραγράφων. Και δεν έκαναν τίποτα άλλο. Τρει παράγραφοι. Έκθεση τριών παραγράφων. Αυτή ήταν η βάση και για νομικέ διαδικασίε. Παρά το ότι είναι εντελώ ανεπαρκή. Οι μαθητέ οι οποίοι εθίγησαν δεν είχαν καμία δυνατότητα διόρθωσης και οποιαδήποτε έφεση για να διορθωθεί η κατάσταση έναντι αυτής της έκθεσης φυσικά απορρίφθηκαν. Πολλά παιδιά λοιπόν είχαν σοβαρό πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά προέκυψαν και το περασμένο καλοκαίρι. Θυμάστε ότι ο Επίτροπος είπε ότι θα γίνει η αναλυτική έκθεση, θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες για να μην ε, ξαναπροκύψουν αυτά τα προβλήματα. Ε, λοιπόν, ξαναπροέκυψαν το περασμένο καλοκαίρι. Με βάση κάποιες εκτιμήσεις, 500 μαθητές ε, είδαν τις δυνατότητες να εγγραφούν σε πανεπιστήμια ε, εν κινδύνου και ορισμένοι δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια. Όλοι οι καθηγητές, όχι κάποιος ακραίος, όλοι οι καθηγητές του Ευρωπαϊκού Σχολείου έγραψαν μία μόνη επιστολή για να υποχρεώσουν να δράσει το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Και είναι σαφής η επιστολή. Σαφής. Παραθέτω λοιπόν από την επιστολή των καθηγητών του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Λένε δεν αναφέρατε ότι εμείς οι καθηγητές που έχουμε πάνω από 100 χρόνια ε, διδασκαλίας χημίας διαμαρτυρόμεθα γιατί ορισμένα θέματα δεν ήταν στην εξεταστέα ύλη ορισμένα θέματα δεν ήταν σαφώς διατυπωμένα υπήρχε υπερβολικά περίπλοκη μαθηματική απέτηση ο τρόπος βαθμολόγησης δεν ήταν συνεπής Νομίζω ότι όταν τα λένε αυτά οι καθηγητές ε, είναι αρκετά ακραία και καταδικαστικά. Και το 12 λοιπόν και το 14 έγιναν σοβαρά λάθη, σοβαρά προβλήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία τα αρνούνται. Δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν την κατάσταση, δεν μαθαίνουν για το μέλλον. Οι μαθητές εξακολουθούν να βλάπτονται ουσιοδός. Όπως είπα, πραγματικά υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις. Ορισμένοι δεν μπόρεσαν να γραφούν στα πανεπιστήμια η κόρη μου μεταξύ αυτών. Μετά από τόσα χρόνια οι καλύτεροι μαθητές μας βλέπουν να θίγονται οι προοπτικές τους λόγω της ανικανότητας των σχολείων, λόγω της ε, γραφειοκρατικής κατάστασης. Παρακαλώ μπορείτε να ολοκληρώσετε, λέει η πρόεδρος. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο και έχουμε πολλούς άλλους ομιλητές. Έχω σχεδόν τελειώσει. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι γίνονται λάθη, αλλά πρέπει να αναμένουμε ότι διορθώνονται. Είναι πολύ σημαντικός ευρωπαϊκός θεσμός. Οι εργαζόμενοι στην Ένωση αναθέτουν την εκπαίδευση των παιδιών του. Δεν διορθώνονται όμω τα λάθη που γίνονται. Το Κοινοβούλιο το 2011 είπε ότι υπήρχε νομικό κενό, είπε ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει σύστημα ανεξάρτητου ελέγχου και τα δικαστήρια και στα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχουν δικαιοδοσία. Τελειώνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το ότι χρηματοδοτεί τα ευρωπαϊκά σχολεία το 2013 300 εκατομμύρια, είπε ότι έχει μόνο μία ψήφο, οι άλλε 28 ψήφοι είναι των κρατών μελών. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα λοιπόν από μόνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δεν το ζητήσετε εσεί, δεν θα γίνει τίποτα υπάρχει ουσιώδες πρόβλημα, θίγονται τα παιδιά μας, το διαπιστώσα το 2011, το είπε το δικαστήριο, το είπε ο διαμεσολαβητής και όμως είναι σαφές ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν εμπίπτουν σε ουσιώδη οικονομικό, συγγνώμη, νομικό έλεγχο και αυτά έθιξαν τα παιδιά μου και άλλα παιδιά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Θεμελιώδεις αλλαγές δεν θα γίνουν αν δεν επιμείνουμε. Θα συνεχιστούν τα προβλήματα και γι' αυτό εγώ υπέβαλα την αναφορά αυτή. Η ζημιά που γίνεται στα παιδιά μας και έγινε στην κόρη μου δεν θα πρέπει να επαναληφθεί και να γίνει και στα δικά σας τα παιδιά. Υπάρχει νομική βάση που πρέπει να αλλάξει για την ίδρυση των ευρωπαϊκών σχολείων. Πρέπει να κατανοήσουμε τα προβλήματα και αυτό ακριβώς είναι που ζητάω στην αναφορά μου. Μια ανεξάρτητη μελέτη δεν μπορεί να είναι κάτι υπερβολικό που ζητάμε. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και ελπίζω να στηρίξετε την αναφορά μου. Πρόεδρος, το 2011 ήμουνα συντονίστρια και στη Νομική Επιτροπή και εισηγήτρια. Ε, συντάκτρια μάλλον γνωμοδότηση στην έκθεση Καβαντά που είχαμε τότε. Το γνωρίζουμε λοιπόν το θέμα. Ναι και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τις λεπτομέρειες σήμερα το βράδυ. Περμολές. Πολύ σύντομα όμως. Γιατί ο συνάδελφός σας πήρε πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόεδρος της Interparants των γονέων. Εγώ είμαι επικεφαλής των ε, γονέων του Ευρωπαϊκού Σχολείου 1. Είχαμε συγκεντρώσει λοιπόν υπογραφές πριν από λίγα χρόνια για να αντιδράσουμε στις ε, περικοπές που γίνονται στα ευρωπαϊκά σχολεία και που οδήγησαν σε μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών σχολείων, βασικά για να γίνουν οικονομίες, χωρίς όμως να γίνει καμιά άλλη σοβαρή ανάλυση. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τρία χρόνια μετά, έχει νόημα η αναφορά αυτή. Η απάντηση είναι πως ναι, έχει. Γιατί, γιατί δεν έγινε καμία αξιολόγηση όσον αφορά την, σε επιπτώσεις της μεταρρύθμισης, δεν έγινε καμία παιδαγωγική ανάλυση όσον αφορά τις αλλαγές αυτές. Και έτσι είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου τα μαθηματικά για παράδειγμα αντί για 6 ώρες γίνονται 4 επειδή ο αριθμός των μαθητών δεν δικαιολογεί να γίνονται όλα τα μαθήματα. Μια άλλη παράδοξη κατάσταση είναι ότι οι τάξεις πρέπει να μπαίνουν μαζί για να μπορούν να καλύψουν τον αριθμό που χρειάζεται και τώρα το κέρδος από όλα αυτά είναι πολύ μικρό. Οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις δεν βοήθησαν να αλλάξει η κατάσταση των ευρωπαϊκών σχολείων. Είμαστε σε ένα σπιράλ προβλημάτων, τα οποία γίνονται όλο και πιο σοβαρά όσο περνάει ο καιρός. Οι χώρες μέλη από την πλευρά τους δεν στέλνουν καθηγητές. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αυξήσει τη δικιά της οικονομική συνεισφορά στα ευρωπαϊκά σχολεία για να μπορέσει να πληρώσει τοπικούς καθηγητές που προσλαμβάνονται. Όλα αυτά έχουν βέβαια επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά έχουν επιπτώσεις και στην παιδαγωγική ισορροπία των σχολείων, γιατί οι καθηγητές αυτοί που προσλαμβάνονται επί τόπου δεν έχουν κανένα σύστημα επιθεώρησης σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τους καθηγητές οι οποίοι στέλνονται από τα κράτη-μέλη που αυτοί ναι επιθεωρούνται. Γίνονται συζητήσεις λοιπόν τώρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε ποιος είναι τελικά αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Η συζήτηση αυτή παρατείνεται. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταλήξει. Πιστεύουμε όμως ότι για τα προβλήματα αυτά που έχουμε από το 2011 δεν μπορούν να λυθούν σαν ένα patchwork, λύνοντας κάποια μικρά προβληματάκια. Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προβλέψει μια γενικότερη επανεξέταση των ευρωπαϊκών σχολείων για να διασφαλιστεί το έργο τους. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Γενικό Κραματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων τώρα για να απαντήσει στα όσα ακούσαμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούσατε δύο ομιλητές που επισήμαναν τα προβλήματα που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά σχολεία. Προφανώς και δεν είμαστε τέλειος οργανισμός και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη, Πήραμε πάρα πολλές ε, συμβουλές, ε, συστάσεις, ε, το Σώμα των Επιθεωρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο και πολλοί άλλοι που είναι αρμόδιοι τα σχολεία μας συσκέπτονται από αυτών των προτάσεων. Θα ήθελα σχετικά με τα νομοθετικά να σας ενημερώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε για την έκθεση που υποβλήθηκε και εξέτασε επίσης και τις συστάσεις του κύριου Κάβερα. Εμείς ε, συστήσαμε μεταξύ άλλων μια νομική επιτροπή η οποία μεταξύ άλλων εξετάζει και την ε, κατάσταση απονομικής κοπιάς που επικρατεί στα ευρωπαϊκά σχολεία. Στην ομάδα εργασίας θα έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαμαρτυριών ε, και θα συζητήσουμε και με πολλούς άλλους αρμόδιους το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στα ευρωπαϊκά σχολεία. Είναι πολύ δύσκολο τώρα ήδη να πούμε ποια είναι η κατάσταση στα ευρωπαϊκά σχολεία. Πάντως ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Τώρα όσον αφορά το ε, νομικό πλαίσιο θα ήθελα να ζητήσω από το νομικό μου σύμβουλο να αναφερθεί με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια στο νομικό μας ε, καθεστώς. Καλησπέρα. Για τα ευρωπαϊκά σχολεία, η αναφορία του 2013 του κ. Ράιαν ε, βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία. Διότι δεν είναι σωστό να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν τηρούν τις αρχές του κοινοτικού δικαίου. Στο σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων υπάρχει ε, ένα σώμα προσφυγής που είναι ένα αυτόνομο σώμα το οποίο εξετάζει τις προσφυγές που φτάνουν εκεί για διοικητικούς λόγους. Και για το σκοπό αυτό βασίζεται το σώμα αυτό και στην ίδια ρύθμιση των ευρωπαϊκών σχολείων αλλά και στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν δικαιοδοσία και υπάρχει συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκές οδηγίες που μπορεί με ένα άμεσα να μην εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά σχολεία. Τα ευρωπαϊκά σχολεία όμως οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές και ως επιτοπλίστων οι προσφυγές που φτάνουν στο σώμα αυτό προσφυγών βασίζονται στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου όπως είναι η ίση μεταχείριση, η διάκριση, η νομιμότητα, η αναλογικότητα, ε, προστασία δικαιωμάτων προκειμένου να υπάρχει μια αποτελεσματική προστασία. Όσον αφορά τώρα την ε, προστασία αυτή τη νομική, ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ατέλειες. Όμως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ανάλυση που έγινε, γιατί ναι μεν κατά το παρελθόν η προστασία αυτή δεν ήταν ε, η γιατί κάποιες δράσεις μπορεί να μην ήταν τέλειες, παρόλα αυτά η... το σώμα αυτό προσφυγών έχει διευρύνει το πεδίο του και ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο σε προσφυγές. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε γιατί έχουμε πέντε λεφτά στη διάθεσή μας ακόμα συνολικά. Όχι μόνο για σας, ε. Με δύο λόγια. Τα ευρωπαϊκά σχολεία και τηρούν τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, αλλά επιπλέον έχουν και τη δικιά τους δικαιοδοσία και τη δικιά τους ρύθμιση με διάφορες δυνατότητες προσφυγών και κατά τα άλλα όταν δεν είναι αρμόδιο το σώμα αυτό, τότε μπορεί ο ενάγων να απευθυνθεί σε εθνικές αρχές. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο νομικό κενό. Μανουέλ Άλτεμερ Μερεγκλίνα τώρα είναι η επόμενη αναφορά για τέτοιου είδου διακρίσει. Πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί τη γνωρίζουμε την αναφορά, δεν χρειάζεται να μας την αναφέρετε από την αρχή. Με δύο λόγια σα παρακαλώ, πείτε μα πώ βλέπετε εσεί τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και θα είμαι πολύ σύντομος. Γνωρίζετε το πρόβλημα λοιπόν. Όλοι το γνωρίζουν. Τόσο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στις απαντήσεις της παραδέχεται ότι πρόκειται για πρόβλημα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εκθέσει από το 2008 το παραδέχεται. Και έπειτα υπάρχει και το γεγονός ότι οι Ισπανοί μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι εκείνοι που πηγαίνουν λιγότερο πίσω στη χώρα τους για να σπουδάσουν. Και αυτό ισχύει γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν κάποιους κανόνες μετατροπής των βαθμών που παίρνουν οι μαθητές στα ευρωπαϊκά σχολεία. Και έτσι μειώνεται το αποτέλεσμα, η απόδοση, και έτσι μειωμένη λαμβάνεται υπόψη για την ε, είσοδο στα πανεπιστήμια. Η Γενική Γραμματεία των Ευρωπαϊκών Σχολείων το ξέρει. Υπάρχουν μελέτες και ξέρουμε ότι υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία ζητούν εισαγωγικέ εξετάσεις και χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά εκεί σε κάποια μαθήματα που δεν έχουν διδαχτεί στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Άρα ήδη εδώ υπάρχει ένα σαφές μειονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι χώρες μέλη είναι οι μόνες που είναι υπεύθυνε για την οργάνωση των εκπαιδευτικών του συστημάτων. Ωραία, συμφωνώ. Αλλά εφόσον τηρούν την αρχή της μη διάκρισης. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Και κάτι ακόμα. Για να πάει κανείς στις εξετάσεις αυτές που δεν είναι μεν υποχρεωτικές, αλλά είναι αναγκαίες αν θέλει κάποιος να σπουδάσει ιατρική ή κάτι άλλο όπου υπάρχει περιορισμένο αριθμός εισακτέων. Οι ημερομηνίε των εξετάσεων αυτών συμπίπτουν με τις ημερομηνίε που οργανώνονται οι εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό Πολιτήριο, το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρέα. Να, παράδεκτη μια τέτοια κατάσταση. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα αυτό με τις Ισπανικές αρχές. Για χρόνια το προσπαθούμε και δεν καταλήξαμε σε λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα, λέει ότι δεν υπάρχει προφανής διάκριση, ενώ για μένα είναι προφανέστατη διάκριση, τόσο στην εφαρμογή της μετατροπής της βαθμολογίας, όσο και στην οργάνωση των εξετάσεων. Τέλος, τα δύο τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα τα πανεπιστήμια μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες που επιθυμούν. Οπότε και εδώ υπάρχει ένα κενό, γιατί τα πανεπιστήμια δεν έχουν υιοθετήσει τους κανόνες και οι μαθητές στα ευρωπαϊκά σχολεία δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Συνόψεις όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ευχαριστώ πολύ. Σολεδάδ και εσείς θέλετε το λόγο από αυτού. Καταρχάς να πω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία θεωρούνται ένα προνόμιο το οποίο γι' αυτό ακριβώς ε, πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερβολικό αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων στην Ένωση είναι μια υπηρεσία, δεν είναι δικαίωμα, είναι αναγκαία υπηρεσία για να μπορούν ε, ορισμένοι να έρθουν και ενδεχομένως για περιορισμένο χρονικό διάστημα Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να πάνε τα παιδιά σε ευρωπαϊκό σχολείο. Δεν είναι λοιπόν προνόμιο. Είναι υπηρεσία. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να προκαλείται διάκριση κατά των μαθητών. Είναι σαφές ότι δεσμεύονται τα διάφορα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν και από ό,τι έχω ακούσει γίνονται περικοπές. Δεσμεύονται και πρέπει να αναγνωρίζουν λοιπόν τα σχολεία αυτά. Βεβαίως στέλνουν και καθηγητές για τα τμήματα τα αντίστοιχα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει όμως σαφής αναγνώριση από τα κράτη-μέλη του εκπαιδευτικού συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων. Οπότε τα παιδιά όχι μόνο φύστανται τις περικοπές που μπορεί να είναι ανησυχητικές, Υφίστανται λοιπόν βέβαια και άλλα παιδιά στις χώρες ε, τις επιπτώσεις των περικοπών, αλλά αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται οι βαθμοί που παίρνουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια της χώρας προέλευσης. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να υπάρξει αυτή η αναγνώριση της βαθμολογίας και να αναγνωρίζεται ισότιμα, ισότιμα να μην γίνονται διακρίσεις για τους μαθητές αυτούς. Πολύ σύντομα. Σωστά είπατε, το 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Παρακαλώ λοιπόν, πρέπει να διαπιστώσουμε τουλάχιστον ότι δεν εφαρμόστηκε αυτό το ψήφισμα. Οι ενδιαφερόμενοι δεν διαπίστωσαν καμία εφαρμογή. Αλλά πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε με το ψήφισμα αυτό έναντι και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Είχα πει τότε, μα το έχετε ξεχάσει, είναι σαν παραμελημένο παιδί. Τα κράτη-μέλη υποτίθεται ασχολούνται. Και τώρα το αφήνουμε, δεν ασχολούμεθα. Να γράψουμε μια επιστολή και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Παρακαλώ εφαρμόστε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, άκουσα τώρα, διάβασα, ότι τα πανεπιστήμια κάνουν ε, τις δικές τους εισαγωγικές εξετάσεις. Τότε να γίνονται για όλους αυτά. Δεν είναι δυνατόν να, ορισμένοι να υποβάλλονται σε αυτές τις εξετάσεις και άλλοι όχι. Και στις επαφές με τις ε, ισπανικές αρχές πρέπει να τονίσουμε εάν υπάρχει ή όχι διάκριση. Εάν υπάρχουν εξετάσεις να υπάρχουν για όλους. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι εσύ που είσαι από αυτό το σχολείο ή από αυτή την περιοχή αναγνωρίζει τη βαθμή σου ενώ άλλον όχι. Λοιπόν, να την αφήσουμε ανοιχτή. Και για το θέμα των Ισπανικών Πανεπιστημίων να ρωτήσουμε πόσο έχουν προχωρήσει οι συζητήσει μεταξύ Κομισιόν και Ισπανίας γιατί η απάντηση της Κομισιόν αφήνει κάποιο περιθώριο ελπίδας ότι αυτές οι διακρίσεις έχουν σχεδόν καταργηθεί. Αλλά δεν καταλάβω πολύ καλά και δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε περαιτέρω. Οπότε παρακαλώ να έχουμε πιο σαφή απάντηση από πλευρά της Ισπανίας. Ευχαριστώ πολύ λέει πρόεδρος. Ξέρετε ότι θα φύγουν οι διερμηνείς σε λίγο. Θα πρότεινα λοιπόν να επανέλθουμε έναντι της Επιτροπής αργότερα για το θέμα αυτό, γιατί διαπιστώνουμε. Βεβαίως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αλλά κάπως ευρύτερα. Να συνεχίσουμε την έκθεση, να, να ζητήσουμε να υπάρξει συνέχεια για την έκθεση Καβαντά και να απευθυνθούμε άλλη μια φορά στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και να ζητήσουμε να μας δώσουν αναλυτική πληροφόρηση για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά βεβαίως να μην βλάπτονται και πρέπει να υπάρχει μία ε, στεναρή νομική βάση. Ο κύριος Μαρτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ οι αναφορές αυτές να μείνουν ανοιχτές και εγώ θέλω να μάθω περισσότερα. Αλλά για την τελευταία παρατήρηση νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω ερμηνεία προθέσεων αλλά θα ήθελα να ξέρω αν είναι μοναδική η περίπτωση του κυρίου ή υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Όταν κάποιοι μαθητές έχουν τελειώσει το Ευρωπαϊκό Σχολείο εάν περνάνε εισαγωγικές εξετάσεις αυτοί είναι οι κανόνες. Να ζητήσουμε στα πανεπιστήμια τη κάθε χώρα να προσαρμοστούν ε, στα ευρωπαϊκά σχολεία. Το αντίστροφο ισχύει. Θα ήθελα να ξέρω αν ε, το διδακτικό πρόγραμμα των ε, ευρωπαϊκών σχολείων είναι κατάλληλο για να μπορεί κανεί να μπει μετά στα πανεπιστήμια. Να έχει δηλαδή ισότιμε ευκαιρίε για να μπει στα πανεπιστήμια να επιτύχει στι αγωγικέ εξετάσει. Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν κάποια στοιχεία. Έχουν προκύψει άλλα τέτοια προβλήματα ή αφορούν μόνο κάποιε περιπτώσει μεμονωμένε. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω αυτή, σε αυτήν την ε, επαφή μας με το Συμβούλιο να αναφερθούμε στην ετερότητα της Ισπανίας. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα ε, εισαγωγής αυτών των συγκεκριμένων μαθητών της Ισπανίας στα πανεπιστήμια. Mr. Kivinen. Ο κύριος Το Ευρωπαϊκό Μπακαλόρεα αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες μέλη και μπαίνουν στα πανεπιστήμια οι μαθητές μας και μάλιστα πολύ καλά. Θα ήταν ενδιαφέρον πράγματι να μελετήσουμε περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικά χρόνια έκανε μία μελέτη που έχουμε στη διάθεσή σας. Το πρόβλημα της Ισπανίας έχει να κάνει με την βαθμολόγηση που είναι 0% και περνάει κανείς αν έχει 60%, ενώ στην Ισπανία περνάει κανείς αν έχει 50%. Οπότε, όντως είναι κάποιοι μαθητές που η βαθμολογία τους μετατρέπεται από τις ισπανικές αρχές και έτσι μένω απ' έξω. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η Ισπανία συμμετέχει στο σύστημα ευρωπαϊκών σχολείων και στο ευρωπαϊκό μπακαλωρεά. Αυτό σημαίνει ότι το δικό μας μπακαλόρα είναι κάπως διαφορετικό από τα εθνικά συστήματα. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει κοινή κατανόηση με την Ισπανία και να βρούμε λύση. Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει φτιάξει μια ομάδα εργασία αξιολόγηση και προσπαθούμε να εξετάσουμε γενικότερα το σύστημα αυτό αξιολόγηση. Την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα εργασία έκανε τι πρώτε προτάσει ζήτησε να μελετήσει λίγο περισσότερο το θέμα για να είναι πιο συγκεκριμένες αυτές και κατά πάσα πιθανότητα θα τροποποιήσουμε το σύστημα βαθμολόγησης για να ε, συνάδει ακόμα περισσότερο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν τέτοιο σύστημα σαν το δικό μας. Πάντως δουλεύουμε πάνω σε αυτή την αλλαγή. Θα ήταν καλό η Ισπανία να σέβεται τις προδιαγραφές μας. Εξαιρετικά. Μάλιστα, προτείνω το εξή σέβομαι απολύτως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι σίγουρη ότι έχετε σημειώσει όλα σε πόθηκαν. Οπότε, ας κάνουμε το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στην Επιτροπή Αναφορών γραπτά, αν έχετε επιπλέον πληροφορίες ή επιπλέον προτάσεις που έχετε να κάνετε γραπτά. Και επιπλέον, όταν η ομάδα αυτή αξιολόγηση, στην οποία αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όταν έχει έτοιμες τις προτάσεις της, στείλτε τες σε εμά στην Επιτροπή Αναφορών. Έτσι θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε όλο το θέμα και θα επανέλθουμε στους αναφέροντες έγκαιρα. Εν ευθέτω χρόνο, όταν θα έχουμε δηλαδή περισσότερα στοιχεία. Συμφωνείτε? Ναι, από ό,τι βλέπω. Καλώς. Δεν είμαι απολύτως πεπισμένη βέβαια ότι αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τι να κάνω, δεν θα έχουμε άλλο διερμηνή, οπότε πρέπει να σταματήσουμε για να συνεχίσουμε με γραπτή διαδικασία. Ε, Ευχαρίστω να επανέλθουμε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο θέμα και είναι πολύ καλό που θα το επανεξετάσετε, όμως υπάρχει ένα σημείο, το σημείο 19, αναφορά της κυρίας Μπάρμπαρα Μαζουργεύσκα Ζαλέσκα 353 του 2011 και 74 υπογραφές όσον αφορά οικονομικές περικοπές στον προπολογισμό. Εγώ ήρθα για να συζητήσω και αυτό το θέμα μαζί σας. Υπήρχε αύξηση 6,5% στον προπολογισμό, δεν υπήρξε μείωση. Υπήρχε αίτηση για 11% αύξηση το Συμβούλιο ή μάλλον οι αρχέ του προπολογισμού μείωσαν την αύξηση αντί για 10% έδωσαν 6,5% αύξηση, αλλά δεν υπήρξαν περικοπέ. Όσον αφορά λοιπόν αυτέ τι αναφορέ για τι οικονομικέ περικοπέ, πολύ θα θέλαμε να κλείσει η διαδικασία επί των δύο αυτών αναφορών. Πρόεδρος. Η αναφορά αυτή είναι μια αναφορά στην οποία απαντήσατε. Όλοι ζούμε σε χρόνους λιτότητας, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να μας δώσετε παραπάνω πληροφορίες έτσι κι αλλιώς. Έχετε επευθυνθεί για μας, μας τα έχετε εξηγήσει. Αλλά θα βάλουμε όλες μαζί αυτές τις αναφορές και θα απαντήσουμε σε όλες αυτές μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την απάντησή σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, Καλό βράδυ. Η μέρα ήταν μεγάλη για όλους μας και φαντάζομαι ότι είσαστε κι εσείς εξαντλημένοι. Αύριο όμως είναι μια νέα μέρα για νέες ευκαιρίες. Καλό βράδυ.